Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start, I'm sure, maybe some more. Κυρίε και κύριοι, αρχίζουμε, ίσω έρθουν και άλλοι, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για να μην καθυστερήσουμε. Κι άλλο. Οπότε με μεγάλη μου τιμή θα συμπροεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση. καλώ ε, όρισε ο επίτροπο ε, κ. Μπρετό ε, και από τι ε, δύο επιτροπές μας η ευχή και θα συμπροεδρεύσουμε με τον συνάδελφο και από την Ήτρε και από την ΙΜΚΟ ε, επομένως και να ξεκινήσω από πλευράς της ΙΜΚΟ ε, θα γνωρίζετε ότι η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε με τις αναδεόμενες τεχνολογίες είναι ατμομηχανές για την οικονομική ανάπτυξη και εννοώ την αυτοματοποιημένη διαδικασία ε, παραγωγής αποφάσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, τα σχετικά με τα μηχανήματα, οπότε και οι επιτροπές μας εννοείται ότι ενδιαφερόμαστε για το τι επιπτώσεις έχουν στην ενιαία αγορά αυτές οι νέες τεχνολογίες, αλλά και τι επιπτώσεις έχουν για τον καταναλωτή. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη και είναι και το θέμα της εναρμόνισης των κανόνων, κανόνες για την αξιοπιστία της παραγωγής και των προϊόντων. Την... Τυποποίηση, βελτίωση των προϊόντων, ε, ενημέρωση για τους καταναλωτές, όλα αυτά είναι σημαντικά αν θέλετε να έχετε εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές και ισότιμους όρους ε, παιχνιδιού για τις επιχειρήσεις. Με αυτά τα σύντομα σχόλια θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο Τιέρη ε, Μπρετών σε αυτή την κοινή μας συνεδρίαση. Θα ακούσουμε τη δική του τοποθέτηση και θα, ακούσουμε, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια όλες τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε φυσικά το διάλογό μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους για περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να σας δώσω τώρα μερικά ε, πρακτικά ε, στοιχεία ενημερωτικά. 15 ε, λεπτά θα μιλήσει ο Επίτροπος και μετά θα έχουμε 14 ερωτήσεις στον πρώτο γύρο από τους συντονιστές ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ όλων των πολιτικών ομάδων. Κάθε συντονιστής θα ρωτήσει για δύο λεπτά και ο Επίτροπος θα απαντήσει ε, για άλλα δύο λεπτά ή τέσσερα. Ξέρω εγώ θα είμαστε ε, σύνολο τέσσερα δηλαδή, ε, αρκετά αυστηροί, γιατί υπάρχει και δεύτερος γύρος 20 ερωτήσεων, αν καταφέρουμε να πάρουμε 20 ερωτήσεις, όπου η ερώτηση θα διαρκεί ένα λεπτό και θα ομαδοποιούμε τις ερωτήσεις ανά 10. 10 ερωτήσεις του ενός λεπτού και θα έχει 5 λεπτά ο Επίτροπος για να απαντήσει στη συνέχεια και όπως καταλαβαίνετε θα ε, κάνει και καταληκτικά σχόλια ο ίδιος ο Επίτροπος και ο συνάδελφος Μπουσόη και θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Παρακαλώ κύριε Επίτροπο, κύριε Βρετό, με ανυπομονησία περιμένουμε να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητά μέλη των Επιτροπών Ήτρε και ΕΜΚΟ. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι έχω την ευκαιρία σήμερα να απευθυνθώ στις δύο επιτροπές. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα για εμάς. Αυτό είπαμε και στο σώμα των επιτρόπων. Έγινε η συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά ήρθα εδώ. Αν μου επιτρέπετε τώρα θα μιλήσω την μητρική μου. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Αλλά βλέπω ότι τα χρειάζεστε όλοι και χαίρομαι ιδιαίτερος. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να περάσω στα γαλλικά και να σας ε, γιατί ε, συζητήσαμε σήμερα το πρωί στο Σώμα των Επιτρόπων, ήταν πάρα πολύ ε, μακρά η συνεδρίαση, Δίρκησε πάρα πολύ, διότι το θέμα που θα μοιραστώ μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται φυσικά για την ψηφιακή μας στρατηγική ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο για τα επόμενα έτη. Είναι τρία ε, τα θέματα τα οποία και από κοινού θα συζητήσουμε. Πρώτον, η στρατηγική μας, η ψηφιακή για τα επόμενα έτη, όπως σας είπα, με ένα φύλλο πορείας οδικό χάρτη πάρα πολύ συγκεκριμένο, με διάφορε διαστάσει και ε, προσεγγίσεις. Το δεύτερον, και είναι πραγματικά αυτό ε, πρωτότυπο καινοφανέ, μια ευρωπαϊκή στρατηγική συντονισμένη για τα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα και γενικότερα τα δεδομένα είναι στην καρδιά της ψηφιακής μετάβασης και θα ε, ταρακουνήσουν ε, την οικονομία μας, τη βιομηχανία μας, την κοινωνία μας. Και το τρίτο είναι μια λευκή βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, για ένα οικοσύστημα αριστείας αλλά κυρίως εμπιστοσύνης η κεντρική ιδέα είναι η εμπιστοσύνη και θα ανοίξει μια μεγάλη διαβούλευση για το επόμενο τρίμηνο ε, για τη Λευκή Βίβλο και ξέρω ότι θα συμμετέχετε και περιμένω πολλά ε, κατά τα άλλα από τις συζητήσεις που θα έχουμε ε, επ' ευκαιρία αυτής της διαβούλευσης. Καταρχάς λοιπόν, η στρατηγική μας για να διαμορφώσουμε το ψηφιακό μέλλον της Υπήρου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι βαθιές οι μεταρρυθμίσεις και ο μετασχηματισμός κυρίως από την ψηφιακή τεχνολογία καθημερινά, την οικονομία μας, τη βιομηχανία μας. Και φυσικά οι τεχνολογίες θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία ε, των πολιτών και όχι το αντίθετο, δηλαδή να είναι πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας και όχι εκπτώσεις με τις νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές, οι οποίες θα πρέπει να αντανακλούν και θα επανέλθω στη συνέχεια στην τεχνητή νοημοσύνη, τις αρχές μας και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είναι πιο ε, ασφαλείς και πιο προσβάσιμες οι διάφορες τεχνολογίες. Μπορώ να αναφερθώ επιμέρους, ε, ας πούμε, για την ε, διάγνωση στην ιατρική, να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα κτλ. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πιο εύκολα να κινούνται και με πάσα ασφάλεια σε αυτό τον ψηφιακό ε, κόσμο, ανεξαρτήτως της ηλικία τους θα πρέπει να προσαρμόζονται και του φίλου φυσικά. Ε, είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι στην ισότητα που θα πρέπει να διαφυλάσσεται ή ακόμα και η επαγγελματική τους ε, διαδρομή. Αυτό που σήμερα όμως σας παρουσιάζουμε και καταπληκτική ευκαιρία για την Ευρώπη για μια βιώσιμη ανάπτυξη για τις εταιρείες μας που χρειάζονται ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να ε, αναδύονται, να αναπτύσσονται, να μοιράζουν όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και να ανταγωνίζονται μια την άλλη, καθώς και να συνεργάζονται επί ίσης όρης που θα έχουν οριστεί ξεκάθαρα. Θέλω να αφαιρθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Πρώτον, τη δυνατότητα της Ευρώπης να γίνει ε, Παγκόσμιο ε, Πρωταθλητή στα ψηφιακά. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να ελέγξει τις βασικές τεχνολογίες και υποδομές. Είναι ένα θέμα τεχνολογικής κυριαρχίας που είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Επίσης, όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, η βιομηχανία θα πρέπει να ασχοληθούν με τις τεχνολογίες, με το 6G, ε, τους υπερυπολογιστές ε, και τα λοιπά. Το ψηφιακό μας πρόγραμμα θα πρέπει να είναι στο ύψος των περιστάσεων και των φιλοδοξιών μας και προσβλέπω σε εσά και υπολογίζω στο Κοινοβούλιο για να ακουστεί η φωνή μας όταν έρθει αυτό το θέμα ενώπιόν σας και ελπίζω να γίνει αυτό. Στη συνέχεια ασφάλεια, η συνεργασία για την ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς και ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε για να βελτιώσουμε ε, τη δυνατότητα να απαντούμε στις επιθέσεις στις ηλεκτρονικές ε, και για τις ε, βασικές υποδομές. Θα τα συζητήσουμε αυτά για την 5G και θα σας προτείνουμε μέχρι το τέλος του έτους μια στρατηγική συνεκτική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και για τις πλατφόρμες, το είπατε πρόεδρε στην εισαγωγή σας, δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε μια κατάσταση όπου ορισμένες πλατφόρμες ε, θέτουν αμφιβόλο και σε κίνδυνο ε, λόγω μιας χαλάρωσης της δημοκρατίας μας, της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Και το λέω ξεκάθαρα. Και το λέω και στους διαχειριστές όταν μας ζητούν ε, να μας δουν όπως έγινε πρόσφατα ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Και για να συνοψίσω θα με έχετε ακούσει να λέω ότι οι πλατφόρμες πλέον θα πρέπει να προσαρμοστούν στην Ευρώπη και όχι η Ευρώπη να προσαρμοστεί σε αυτές. Και φυσικά προς την κατεύθυνση αυτή θα δράσουμε. Άρα, έχουμε την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που προετοιμάζουμε για το τέλος του έτους, για πιο σαφείς ε, αρμοδιότητες και ευθύνες ε, αυτών των πλατφορμών. Όπως είπατε και ε, για κάποιο περιεχόμενο τελείως απαράδεκτο που φιλοξενούν. Επίσης, όλο και περισσότερο θα κοιτάξουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια εκ των προτέρων ε, ρύθμιση, νομοθέτηση, όπως κάναμε για την αγορά των τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ελέγχουμε και εδώ ε, σας μιλώ φυσικά ως Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, να ελέγχουμε το μερίδιο της αγοράς και την εξουσία που έχουν κάποιες πλατφόρμες που έχουν γίνει ε, ε, ρυθμιστές, ας πούμε, gatekeepers ε, ουσιαστικά, απόλυτοι και δεν γίνεται αυτό για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έρχομαι τώρα στη στρατηγική για τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν νοείται τεχνητή νοημοσύνη χωρίς δεδομένα. Άρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα στο σκεπτικό μας. Την τελευταία δεκαετία είδαμε όλοι τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα δεδομένα και ε, κυρίως τα προσωπικά δεδομένα. Γεννήθηκαν διάφορες πλατφόρμες, τα έχουμε δει όλοι αυτά, όχι στην Ευρώπη. Και συχνά ανησυχούσαμε και σωστά ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες φυσικά και στην Κίνα. Και θέλω να σα το πω απλούστατα χωρίς καμία αλαζονία και ε, πολύ ταπεινά. Πριν από 10, 12, 14 χρόνια ξεκίνησαν αυτές οι πλατφόρμες και αυτό δεν ήταν καμιά τρομερά περίπλοκη τεχνολογία και εδώ σας το λέω ως μηχανικός. Ε, δεν ήταν κβαντικοί υπολογιστέ αυτές οι πλατφόρμες, ήταν μια στοιχειώδης τεχνολογία βασική που υπήρχε τότε, συναρμολογήθηκε, ε, αγόρασαν ε, κάποια επιμέρου στοιχεία και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν. Φυσικά γιατί υπήρξε άμεση πρόσβαση, ευρύτατη και με πολύ μεγάλο πελατολόγιο που δημιουργούσαν δεδομένα και προσωπικά δεδομένα τα οποία ε, ρούφηξαν αυτές οι πλατφόρμες ε, με αμφισβητούμενους όρους πολλές φορές ε, και μπράβο στο Κοινοβούλιο γιατί είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε και ήταν ε, σωστό να ρυθμιστούν και σιγά σιγά έγινε και στην Κίνα και άρχισαν να ξεφυτρώνουν αυτές οι πλατφόρμες και ε, σκεφτήκαμε, θεωρήσαμε ότι κάπου είχαμε χάσει τη μάχη. Και πραγματικά το λέω αυτό ταπεινά. Για ποια είναι αυτή η φάση. Πριν από 10-12 χρόνια, όχι πριν από 50 χρόνια, είναι πρόσφατη αυτή η εξέλιξη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή γιατί αλλάζει ε, πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και καταναλώνουμε και έχουμε και κάποιο συστημικό αντίκτυπο ε, στα δημοκρατικά μας δικαιώματα και καλούμαστε να δράσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Το είπαμε όμως ότι έχουμε ένα νέο κύμα το οποίο επίκειται με τα δεδομένα που δεν είναι πλέον προσωπικά κατά κύριο λόγο, αλλά είναι δεδομένα ε, βιομηχανικά. Με την ευρία έννοια παρακαλώ να το εκλάβετε αυτό. Ε, στο 5G, όλα αυτά τα διασυνδεδεμένα αντικείμενα, ε, το ονομάζουμε το διαδίκτυο ε, των ε, αντικειμένων, μέχρι το 2020 θα έχουμε 500 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια επαναλαμβάνω, στον πλανήτη αντικειμένων που θα είναι διασυνδεδεμένα και θα αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ως προς τα δεδομένα. Το ίδιο ισχύει για τα digital twin ε, στη βιομηχανία, για τα αυτοκίνητα, για την υγεία, για την κινητικότητα, σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όλα αυτά γίνονται από το δίκτυο 5G. Θα αναφερθούμε σε αυτό στη συνέχεια, αν θέλετε. Σήμερα, λοιπόν, τελειώνει αυτό το κύμα, μάλλον αρχίζει τώρα απέναντί μας αυτό το τεράστιο κύμα των ε, δεδομένων και το έχω πει επανελειμμένα, από καταβολής κόσμου, μέσα σε 18 μήνες ε, θα ε, παράξουμε ε, ό,τι έχουμε παράξει από την αρχή της ανθρωπότητας, 43 εκατομμύρια δεδομένα. Και η Ευρώπη δεν έχει απλώς ένα ρόλο να παίξει, αλλά πολύ σημαντικό και δεν έχει καθυστερήσει, γιατί είναι η πιο ε, αναπτυγμένη η βιομηχανική μας βάση και αυτά τα δεδομένα θα ε, προέλθουν από τη βιομηχανική βάση και την εκμετάλλευση των νέων εξελίξεων και των νέων τεχνολογιών, όπως σας είπα. Από το δίκτυο 5G και τις αντίστοιχε υπηρεσίες. Και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά εδώ θα πρέπει να έχουμε τις υποδομές που χρειάζονται, δεν υπάρχουν ακόμα. Μία προσωπική πλατφόρμα ε, είναι περίπλοκη, αλλά όχι πάρα πολύ. Μία βιομηχανική πλατφόρμα για βιομηχά δεδομένα είναι πολύ πιο βαριά, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και στην Ευρώπη θέλουμε να αναπτύξουμε σε όλη την Ήπειρο την ασφάλεια για να βοηθάει και τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τις εταιρείε μας και τις επιχειρήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δαπανίσει μέχρι 2 δισεκατομμύρια ευρώ για ε, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και βιομηχανικά cloud ε, ε, για ένα, ένα δημόσιο πυλώνα και έναν ιδιωτικό πυλώνα cloud to edge θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό το σχήμα. Υπάρχει ήδη για πιο δημόσια δεδομένα θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε ακριβώς ε, για ε, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, το τρίτο στοιχείο είναι ε, η ε, Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί ήσασταν πάρα πολύ δραστηροί, μας ε, βοήθησαν πάρα πολύ τα έγγραφά σας, έγινε πολύ μεγάλη δουλειά και ήταν πηγή έμπνευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αρχίσουμε να προχωρούμε προς τη φάση της ευρεία διαβούλευσης για τη Λευκή Βίβλο. Πραγματικά αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια δομή που θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη στους πολίτες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Υπάρχει αγωνία, φόβος, άγχος, όλα αυτά είναι θεμητά. Τι θα γίνει με τους αλγορίθμους, ποια χρήση θα γίνεται. Φυσικά οι αλγόριθμοι αυτοί θα πρέπει να αντανακλούν ε, όλες τις αρχές και αξίες που χρόνο με το χρόνο έχτισαν την Ευρώπη μας. Ηθικές, δεδολογικές αξίες, διάφορες ε, ε, ε, υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων, όλα αυτά θα πρέπει να αντανακλώνονται και στους αλγορίθμους. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χρήση. Να δούμε αν ε, ε, ε, υπάρχει κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο, πολύ συγκεκριμένα να μελετήσουμε. Είναι μεγάλο διακύβευμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Α πούμε στην ιατρική όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που ε, βοηθάει ένα χειρουργό να κάνει μια εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. είναι πολύ κρίσιμη αυτή. Ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, ποιο αλγόριθμο έτσι ώστε να είναι συμβατά και με τον άνθρωπο. Ε, είναι κλεμμένα αυτά τα στοιχεία, έχουν υπολογιστεί, έχουν ενέχουν τις αξίες και τις διαφορές μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι ε, που χρειάζονται έλεγχο στην Ευρώπη. Μπορούν να έρθουν και άλλες εταιρείες από αλλά ε, θα πρέπει να έχουμε και λόγο. Υπάρχουν και άλλοι αλγόριθμοι που είναι λιγότερο κρίσιμοι ή αμφισβητούμενοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε προτάσεις ε, για επισήμανση, ακριβώς για να ξέρουμε τι περιέχει ο κάθε αλγόριθμος. Είναι πολλές οι περιπτώσεις και αντίστοιχες ή ε, δράσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη ε, διαβούλευση. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, εκ των προτέρων νομοθέτηση είναι πολύ σημαντικό. Στο τέλος, αν θέλουμε να νομοθετήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε για να έχουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό, ένα πλαίσιο ε, που θα ρυθμίζουμε όπου χρειάζεται σε συνεργασία μαζί σας όλα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, μου δώσατε 15 λεπτά, σας δίνω 15 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Πρώτος είναι ο κύριος Σβάμπ, συντονιστής του ΕΛΚ στην ΕΜΚΟ. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΚ χαιρετίζει την ολιστική και φιλόδοξη πρόταση της ε, Κομισιόν για τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι σωστά αναφέρεται ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην ε, ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι χρησιμοποιούμε τις διάφορες συσκευές, αλλά φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη χάθηκε τα τελευταία χρόνια. Αν δούμε μάλιστα το εύρος των προτάσεων που ε, υποβάλλει σήμερα η Κομισιόν, πάρα πολλά από αυτά έχουν στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από αυτήν την τεχνολογική μεταστροφή ε, θα πρέπει να μπορεί να αντλήσει ένα οικονομικό όφελος για όλους νέους εργαζόμενους εργοδότες επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει νομίζω να ακολουθήσουμε ούτε τον Κίνα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, ούτε της είπα. Πρέπει να επιλέξουμε τον τρίτο δρόμο ε, που θα βασίζεται στις δικές μας θεμελιώδεις αρχές. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε δύο-τρία στοιχεία από αυτά τα οποία είπατε. Είναι σωστό το θέμα των χρηστών να υπάρξει μια ρύθμιση εξ γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού μας δίνει την δυνατότητα να παρέμβουμε εξ πόστο αλλά ε, πλέον είναι τόσο μεγάλη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ώστε όσο ανταγωνιστικές και να ήταν οι ευρωπαϊκές εταιρείε δεν έχουν πλέον καμία ελπίδα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει οικονομικό όφελος και ταυτόχρονα να αποκαταστήσει την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών στην ε, τεχνολογία. Και επειδή είστε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξή Πώς θα καταφέρουμε η εσωτερική αγορά να έχει την μορφή της ε, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία και στα 27 κράτη με την καινοτομία, με τη σκληρή εργασία να μπορέσουν να ωφεληθούν διασυνοριακά να παραμείνουν ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι και ψηφιακά και στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Κύριε Μπρετό. Σας ευχαριστώ κύριε Ανδρέας. Σβάμπ για την ερώτησή σας. Πρώτα πρώτα, το θέμα της εμπιστοσύνης. Ακριβώς αυτό είναι ο στόχος μας, ένα τέτοιο πλαίσιο εμπιστοσύνης. Τώρα παρακάτω όμως δεν πρόκειται εδώ για μια νομοθεσία πριν έχουμε τις εφαρμογές, γιατί αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Να πούμε ότι θα ε, νομοθετήσουμε εκ των προτέρων, αλλά δεν γίνεται αυτό. Ήδη έχουμε κάποιες εφαρμογές και για αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά τα δύο σκέλη. Πρώτα-πρώτα τα προσωπικά δεδομένα και τους ε, αλγορίθμους που βγαίνουν σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά υπάρχουν σήμερα. Σας είπα τι έγινε και για την υστέρηση, οπότε γι' αυτό πρόκειται να γίνει αυτή η πιστοποίηση που θα καλύψει τους πάντες χωρίς ε, διακρίσεις και να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε τον κίνδυνο. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι ό,τι αφορά τον ιδιωτικό βίο, τα προσωπικά δεδομένα, θα ε, ληφθεί υπόψη για αυτούς τους χαλόρυθμους. Και δεύτερον, το δεύτερο κύμα που μιλήσαμε για το πλεονέκτημα, το οποίο ε, αφορά την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη, γι' αυτό και είπαμε ότι ξεκινάει τώρα πόλεμος. Εδώ, εδώ είναι το πρώτο πεδίο της μάχης ε, και όλοι εδώ θα θέλουν να έρθουν και αυτό θα ωφελήσει φυσικά τις επιχειρήσεις μας που θα έχουν την προτεραιότητα και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτό το Data Act, αυτό το ειδικό νομοθέτημα ούτω ώστε ανακλάδο, ανατομέα, αναλυσίδα αξίας από αεροναυπηγική, από αυτοκινητοβιομηχανία, από φαρμακοβιομηχανία ή χρηματοοικονομικά και να έχουμε την πλατφόρμα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι διασυνοριακό. Οπότε έτσι έχουμε αυτή την καινούργια κοινή αγορά των δεδομένων για την βιομηχανία, κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Λάβουμε υπόψη μόνο τα προσωπικά δεδομένα και την πολιτιστική μας πολυμορφία, γιατί αυτό είναι σήμερα το ατού μας. Ή ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Μπρετών. Κρίστιαν Έιλερ. Συντονιστής. ΕΛΚ Ήτρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα έχετε την στήριξη του ΕΛΚ. Υποσχεθήκατε μια φιλόδοξη προσέγγιση και πράγματι αυτό κάνατε. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο στο διοργανικό πλαίσιο και τα επόμενα χρόνια. Πρακτικά μιλώντας, αυτό το οποίο θα πρέπει να επιτυχθεί είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτό είναι στα χέρια μας, μετά είναι το θέμα του προϋπολογισμού και βεβαίως ε, το θέμα του κατά πόσον θα το δεχτούν ε, τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε φιλοδοξίες πρέπει ε, δούμε τελείω διαφορετικά τα πράγματα στο διοργανικό πλαίσιο φέτο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Μιλήστε για μια στρατηγική δεδομένα, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε με τα δικά μα δεδομένα ε, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Και βεβαίω ε, οι θέσει κομισιών ήταν ανοιχτέ και τώρα μαθαίνουμε ότι ίσω υπάρξει κάποια μικρή διαφοροποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε τα τρία θεσμικά όργανα για να ανταποκριθούμε στις ε, συνθήκες. Ε, το ίδιο και με τον ε, προϋπολογισμό. Είναι μικρός ο προϋπολογισμός. Μετά υπάρχει το κομμάτι που είπατε, το κομμάτι το οποίο αφορά την έρευνα για την ασφάλεια. Αλλά πρακτικά έχουμε τις σωστές προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλά νέα σχέδια, αλλά δεν υπάρχει νέο χρήμα. Βεβαίω αυτό αφορά και το πώς ε, τα κράτη-μέλη είναι σε επαφή μεταξύ τους ε, στο ΠΔΠ για να υπάρχει και ο ανάλογος προϋπολογισμός. Γιατί βεβαίως ε, χρειαζόμαστε τον προπολογισμό να πολλαπλασιαστεί. Τα θέλει και ο κύριο Τίμπερμανς μετά για τη Green Deal. Λοιπόν, τι θα γίνει δύο οργανικά και μέχρι το τέλος του έτους. Σας ευχαριστώ κύριε Έλερ, κύριε Λεμπρετό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Έλερ. Ναι, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, οι πόροι για να καλυφθεί η φιλόδοξη προοπτική αυτή, ακριβώς όπως τα είπατε. Πρώτα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή η προοπτική. Είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε πεπισμένοι και έχουμε τον τρόπο ούτω ώστε να είμαστε ενεργοί, να είμαστε δυναμικοί σε σχέση με αυτό το νέο κύμα, να μην είμαστε ουραγοί. Και σας το λέω ειλικρινά, επί τη βάση της πραγματικότητας, της πραγματικής αγοράς, της πραγματικής οικονομίας και βιομηχανίας. Το ξέρω το θέμα. Θα πρέπει βεβαίως να έχουμε τα μέσα προς τούτο. για να περιχαρακώσουμε, να, να έχουμε αυτές τις ανοιχτές πλατφόρμες, αλλά με ασφάλεια των δεδομένων. Μιλάμε για ένα δις γιατί θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες. Δεν έχουμε ακόμα τις απαντήσεις τη λύση. Αλλά υπάρχουν οι προγράμματα και από εκεί θα τα εκταμιεύσουμε. Οπότε και εσείς θα μας βοηθήσετε σε σχέση με τον υπολογισμό, αυτόν ο οποίος τώρα βρίσκεται υπό συζήτηση χωρίς ε, περικοπές. Και αυτό θα διακυβευτεί αμέσως επόμενες μέρες. Είπαμε για αυτή την διτή, διπλή τεχνολογία, αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε, την κβαντική ε, κωδικοποίηση ή κρυπτολογία, όπως τη λένε. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι ήδη όπως είναι σήμερα τα πράγματα πάμε για δύο εκατομμύρια εκταμείευσης. Σχάλτε μόζε. Είναι η συντονίστρια. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρετόν και σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε τα οποία οπωσδήποτε δημιουργούν διάφορες σκέψεις δεν έχω διαβάσει ολόκληρη την Λευκή Βίβλο, αλλά είναι θετικό το ότι έχουμε τόσο νωρίς τόσο μεγάλα οράματα και τόσο μεγάλες σκέψεις και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ισχυρή ε, στα ψηφιακά μέχρι εδώ καλά. Αλλά βεβαίως ως σοσιαλδημοκράτης ε, έχω και κάποια ανησυχία. Λοιπόν, ε, τώρα κάποιες ερωτήσεις. Ε, η Κομισιόν εστιάζει στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Αλλά... Πώς ε, θα μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι τελικά αυτό ο μετασχηματισμός δεν θα οδηγήσει σε μια απορρίθμιση της αγοράς εις βάρος ε, των εργαζομένων ε, και των χρηστών. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης μια συνοχή στην εσωτερική αγορά. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν φοβάστε τη ρύθμιση αν αυτή απαιτηθεί, αλλά... θα τα ζήσουμε αυτά, θα τα νιώσουμε. Πόσο όμως θα τα δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμοί κτλ. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις και εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ε, αναμένουμε ακριβώ να δούμε πώς θα γίνει αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρετών. Ε. Ευχαριστώ, κύριε Σαλντεμόζε, για την ερώτησή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί τη συζητήσαμε σε βάθος. Ε, αυτή η κοινωνική πτυχή, η πλαισίωση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, αυτού του προγράμματος. Έχετε δίκιο. Αυτή η επικείμενη εξέλιξη δεν θα γίνει σε δύο χρόνια. Ε, είναι μακράς πνοής και πολύ βαθιά. Ε, έχουμε όμως και το χρόνο, αλλά και το καθήκον να προετοιμαστούμε αμέσως, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας πίσω και να υποφεληθούν όλοι. Ε, ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας απασχολεί πολύ, και το αναφέρατε κι εσείς, να αποφευθεί ο κίνδυνος απορρίθμισης της εσωτερικής αγοράς. Ποια είναι σήμερα η ισχύ και η ενότητα της ενιαίας αγοράς. Ακριβώς όλα αυτά που κάναμε από κοινού. Ε, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα. Ε, ορισμένοι ε, τα επικρίνουν και κάποιοι άλλοι αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το λόγο. Αλλά αυτή είναι η ισχύ μας. Και τώρα δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να ξυλώνουμε ότι έχουμε οικοδομήσει. Και ε, πραγματικά είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο ιστός οι πλατφόρμες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι το αντίστροφο, ιδιαίτερα οι πλατφόρμες που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες. Και τελικά αυτοί που απασχολούνται είναι μισθωτοί, είναι αυταπασχολούμενοι με όλη την επισφάλεια που ενέχει αυτή η ε, εργασιακή σχέση και πραγματικά μας απασχολεί και γι' αυτό και προτείνουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εναρμονισμένο προφανώς, γιατί η έλευση όλων αυτών των ε, πλατφορμών θα μας επιτρέψει, αν δουλέψουμε καλά, να επιταχύνουμε την εσωτερική αγορά και όχι να την γκρεμίσουμε. Πάντα ε, διαφυλάσσοντας όλες μας τις αξίες. Ευχαριστώ κύριε Μπετού. Η κυρία Τόγια, παρακαλώ, συντονίστρια Ήτρε από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Πάρα πολύ κύριε Παδίου, να σας πω ότι πάρα πολύ χαιρόμαστε για αυτά που είπατε στον ε, Ζούκερμπεργκ. Ήταν ξεκάθαρο τα όσα είπατε, απε, απερίφραστα, χωρίς μισόλογα. Γιατί υπάρχουν τα θέματα τα νομικά, τα θέματα τα φορολογικά και όλοι θα πρέπει, από όπου να είναι, θα πρέπει να αναλάβουν τις ε, ευθύνες τους και κυρίως ε, αυτά που είπατε για τα φορολογικά. Τώρα εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Η Ευρώπη μπορεί και θα μπορεί να έχει μια, ε, ένα νομοθετικό ε, πλαίσιο για την ελευθερία όλων αυτών των κινήσεων αλλά το, το πνεύμα της στρατηγικής σας είναι το να περάσουμε σε αυτή την φάση των μεγάλων επενδύσεων να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά τον ψηφιακό τομέα και ε, οι περισσότερες από τις σημαντικές ε, υποδομές και όσον αφορά τη διαχείριση των ε, δεδομένων είναι βιομηχανικά προϊόντα που φτιάχνονται εκτός Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει προς τα εκεί να στραφούμε. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα. Οπότε και εγώ σας ερωτώ να μου πείτε το ότι θέλουμε τώρα, όπως είπατε, να οικοδομήσουμε κάποιο είδους καταπίστευμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό είναι μια προοπτική που όμως ε, είναι κάτι το οποίο θα, θα περιχαρακώσει, θα περιορίσει τις ε, κρατικές υποδομές γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ε, κέντρο κατευθυνόμενες δομές ελέγχου. Και τι θα γίνει, πώς θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα για υγεία, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Όμως θα πρέπει να έχει κεντρική, πρωταγωνιστική θέση σε όλα αυτά ο πολίτης. Υπάρχει τεχνολογία για να υπάρχει διαλειτουργικότητα, ε, υπάρχει ανωνυμία, Οπότε θα πρέπει αυτό το άρμα να έχει και δημοκρατικό χαρακτήρα. Απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Τόια για την ερώτησή σας. Πάρα πολύ σημαντική φυσικά επίσης. Εδώ υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό εκ των όνου Κάνευ είναι να μπορούν να έχουν πρόσβαση όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δημόσια δεδομένα είναι τεράστια δεξαμενή. Ορισμένα φυσικά πρέπει να μείνουν απόρριτα, ανώνυμα, ε, ανωνυμοποιημένα, αλλά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεών μας, των νεοφυών επιχειρήσεων, των ε, ε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί είναι ένα ε, καταπληκτικό κοίτασμα ε, προόδου και δημιουργίας. Αλλά πέρα από αυτά τα κοινά δεδομένα που θα μοιραζόμαστε όλοι, ας πούμε, στην αυτοκινητοβιομηχανία η βιομηχανική παραγωγή παράγει δεδομένα. Ορισμένα είναι πάρα πολύ απόρριτα γιατί ε, αφορά διπλώματα τεχνίας, ε, εμπορικό απόρριτο. Υπάρχουν κάποια άλλα που μπορούν να τα μοιράζονται και με τους ανταγωνιστές τους. Ας πούμε δεδομένα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση. Ε, όλοι έχουν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα και μπορούν αυτά να συνενώνονται σε κάποιες δομές από δομές διακυβέρνησης που που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση που θα σας ε, καταθέσουμε διακυβέρνηση και ε, νομοθέτηση. Φυσικά όχι δεσμευτική, αλλά ε, ισχυρές ενδείξεις για τη βιομηχανία και για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως σας είπα. Είπατε επίσης ότι χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, φυσικά, και μεγάλα έργα. Προηγουμένως αναφέρθηκα σε αυτά που προτίθεμεθα να κάνουμε. Στο Euro HPC, Είναι και μια δομή αυτή που συνενώνει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε να ενώσουμε την υπολογιστική μας ισχύ με ένα ειδικό cloud που θα προτείνουμε, ένα υπολογιστικό ενέφος για να αποθηκεύονται εκεί τα δημόσια δεδομένα και να μπορούν όλοι να τα μοιράζονται και μετά Ε, ε, θα είναι ευρωπαϊκά αυτά τα project ε, των υπερυπολογιστών και όχι εθνικά. Ο συντονιστής ΕΜΚΟ την Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την δουλειά που κάνατε και για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσω στην δανέζικη γλώσσα. Κοιτάξτε, ο στόχος μας, η αφετηρία μας, αν θέλετε, είναι το ότι η ομάδα μας, ε, η Renew, είναι πάρα πολύ θετική απέναντι σε αυτήν την προσέγγιση. Χαιρόμαστε για το ότι η Κομισιόν επιδεικνύει μια φιλοδοξία. Και έχουμε εκφράσει επίσης ε, την απόψή μας ε, σχετικά η συνάδελφος ε, Σχάλντε Μόζε από τους σοσιαλδημοκράτες θα ήθελε να αποφύγει την απορρίθμιση. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ρωτήσω το εξής. Πώς όμως θα πρέπει να προσέξουμε το τι γίνεται και με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βεβαίως είναι πρωτοποριακός και έχει καθορίσει τι προδιαγραφέ για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, τι μη κερδοσκοπικές. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επιβαρυνθούν ε, υπερβολικά από όλους αυτούς τους κανόνες, αλλά θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Μπρεθόν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λόκεγκάρτ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα μόνο να σας πω ε, εισαγωγικά πριν αρχίσω την απάντησή μου το εξής. Προσπαθώ να ε, μιλώ με γεγονότα και να ε, αγωνίζομαι κατά των fake news, όλες αυτές τις ψευδείς ειδήσει που κυκλοφορούν για την τεχνολογική Ευρώπη, την αδύναμη Ευρώπη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Εγώ από αυτόν τον κόσμο προέρχομαι και σας λέω ότι είναι λάθος όλο αυτό. Και θέλω μαζί με εσά και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν είναι γεγονός αυτό που διαδίδεται ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει. Θα δούμε από κοινού. Φυσικά όλοι θα πρέπει να υποφελούνται και φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα δεν είναι να βαρύνουμε τη γραφειοκρατία για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ο γενικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα και υποφέρουν κάποιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα αυτού του κανονισμού, αλλά να υπάρχουν δομές πιο ευέλικτες, αμοιβιοποιημένες για τις ε, μικρομεσαίες, γιατί είναι πολύ δύσκολη και βαριά η τήρηση. Θα πρέπει όλοι να υποφελούνται από την ίδια προστασία και οι εργαζόμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την προστασία των δεδομένων τους, των προσωπικών, αλλά να μπορέσουν αυτές εταιρείε να επωφεληθούν από αυτό που είναι ισχύς και όχι βραχνά σε τελική ανάλυση και να υποφελούνται όλοι από αυτές τις δραστηριότητε. Γι' αυτό ε, ε, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργάζονται ε, σε κλαδικό επίπεδο, σε αλυσίδες παραγωγής αξίας και όλοι οι αλγόριθμοι που θα επιτρέψουν να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα, θα πρέπει να είναι προς όφελος όλης της αλυσίδας δημιουργίας αξίας. Και έτσι σιγά σιγά φτιάχνουμε δομές εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμοσύνης για να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες να συμμετέχουν. Είμαστε πλήρως λοιπόν ευθυγραμμισμένοι με το δικό σας όραμα και θεώρηση και πιστέψτε με, άκουσα πολλά από όσα είπαν πολλοί από εσά ότι είναι πολύ βαριές οι δικασίες και ε, συμφωνώ, ξέρω, σας γνωρίζω ότι ασπάζεστε αυτές τις αξίες, αλλά και στη χώρα σας βλέπετε ότι κάποιοι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτό το γενικό κανονισμό, ίσως ε, συνεργαζόμενοι με άλλες επιχειρήσεις να τα καταφέρουν καλύτερα η κυρία Μαρτίνα Τλαμπάιοβα από την ομάδα Renew, συντονίστρια στην Ήτρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, βλέπω ότι χαίρεστε. Ε, είστε έτσι ευτυχείς, ε, μας λέτε κάτι συγκεκριμένο, το ποιο είναι το όραμα για το ψηφιακό, το όραμα για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Αλλά η δύσκολη δουλειά μας περιμένει ακόμα. Πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή προπολογισμό την στήριξη των κρατών μελών για το όραμά σας και θα ήθελα να μάθω τι στρατηγική έχετε γι' αυτό. Το να γίνουν σωστές αξιολογήσεις αντικτύπου και να προτείνετε νομοθεσία μόνο όταν αυτή χρειάζεται. Να μην υπάρχει δηλαδή υπερβολική ρύθμιση. Τύπωσα εγώ όλα τα έγγραφά σας εδώ, πάρα πολύ ωραία. Θα τα διαβάσω μετά στο αεροπλάνο και μετά που θα κοιμάμαι. Είμαι σίγουρος όλοι το ίδιο θα κάνουμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ε, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο για τα ζητήματα δεδομένων σε σχέση με τη βιομηχανική στρατηγική. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα αναπτύξουμε στην Ευρώπη τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες των βιομηχανικών δεδομένων. Και ξέρετε, η καιρή τι. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε γρήγορα, να μου πείτε αύριο αυτό, μεθαύριο αυτό θα κάνουμε. Συγκεκριμένα βήματα γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ε, όταν μιλάμε επίσης για τις ε, σχετικές ευκαιρίες για τα βιομηχανικά δεδομένα, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εξίσωση αυτή. Έχουμε κάποιες μικροδιαφορές, ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ, αλλά όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε. Ξέρουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε τις γενικολογίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παράγουν δεδομένα, εκμεταλλεύονται δεδομένα δουλεύουμε δεδομένα και ίσως κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν επιχειρήσεις ε, του δισεκατομμυρίου. Οπότε σας ερωτώ πώς διασφαλίζουμε ότι όλο και περισσότερες ε, επιχειρήσεις θα είναι ε, επιτυχής. Συγκεκριμένα πράγματα πείτε μου. Ένα, δύο, τρία. Αύριο τι θα κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Μπρετών. Με ευχαριστώ. Κυρία Κλαμπάγιοβα για την ερώτησή σας. Ελπίζω να διαβάσετε με χαρά το έγγραφο αυτό και να το διαβάσετε πριν κοιμηθείτε. Ελπίζω να μην σας ε, να νουρίσει, <laughs> αλλά να ε, σας κρατήσει σε εγρήγορση. Είναι λίγο πυκνό το κείμενο, το αναγνωρίζω. Αλλά υπάρχει εδώ κάτι κατεπήγον που απαιτεί να δράσουμε. Αυτό που μας είπατε ε, απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη σε διάφορους βαθμούς και κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και είναι σημαντικό και επίκαιρο γιατί τώρα ε, γίνεται η συζήτηση για τον προπολογισμό. Υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίε και πολλές πολύ πλούσιες ε, και αποδίδουν στα κράτη-μέλη και θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη στρατηγική. Και πιστέψτε με, ε, συμπεριλαμβάνονται, γιατί αυτή είναι η κανονική εξέλιξη του βιομηχανικού κόσμου και του κόσμου των δεδομένων. Φυσικά χρειάζονται πόροι και φυσικά ποντάρουμε σε εσά και υπολογίζουμε σε εσά για τον προπολογισμό, ιδιαίτερα ε, για τα ψηφιακά ε, θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση. Επειδή θέλετε συγκεκριμένες φάσεις, πρώτη συγκεκριμένη φάση, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, η πλατφόρμα για τον Ευρωπαϊκό Υπερυπολογιστή EuroHPC. Έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε από τώρα να το λανσάρουμε για να υπάρξει και ε, αυτή η δυνατότητα που δεν θα είναι μόνο εξαγγελτική θα δημιουργήσουμε έτσι τα πρώτα ε, τουβλάκια, ας πούμε, στα πλαίσια ε, αυτού του υπερυπολογιστή για να τα εκμεταλλευτούμε ε, στη συνέχεια. Ελπίζω η δεύτερη φάση να είναι στο τέλη του έτους ή αρχές του επομένου. Αυτή τη συμμαχία, γιατί θα πρέπει όλοι να οργανωθούν, να συνασπιστούν και ελπίζω πάρα πολύ ένα κλάσμα του προπολογισμού να αφιερωθεί εκεί και ξέρουμε που θα τα βρούμε. Αν αγωνιστούμε από κοινού και θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα είναι πολύ αργά. Αν υπάρχουν και άλλοι ήπειροι στο, μετα... μεταξύ, ε, να συμφωνήσουν μαζί μας, γιατί είναι πάρα πολύ στρατηγικό. Εκεί θα δημιουργήσουμε τους αλγορίθμους για τις βελτιώσεις που θα ε, είναι προς όφελος όλων και όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας και στις μικρομεσαίες, στις οποίες τόσο είστε προσιλωμένοι όπως και εγώ. Ευχαριστούμε, λέει πρώτος και τώρα ο Γιώργος Παύλο Μπόρκια, ο συντονιστής ε, στην Ήτρε η ψηφιακή τεχνολογία στο μέλλον ε, θα γίνει κάτι σαν ψυχρός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και των άλλων εμπορικών ε, δυνάμεων και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις τηλεπικοινωνίες Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνουν τα κράτη-μέλη τα τελευταία 20 χρόνια Είδαμε τι έγινε με τους γίγαντες ε, του διαδικτύου που άλλαξαν το ψηφιακό σύμπαν, οπότε ε, εσείς μας ε, περιγράψατε ποια προσέγγιση προτιμάτε και είδαμε και αυτό το οποίο φασίστηκε για το Facebook. Οπότε αυτή η επανεκκίνηση για την ψηφιακή τεχνολογία θα καθρεφτίζει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις και αναλαμβάνετε την ευθύνη να χρησιμοποιήσετε κάποια μέσα πολιτικής που θα μας προστατεύσουν από πλευράς ψηφιακής. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορέσουν να κοντράρουν τους γίγαντες του διαδικτύου του υπολείπου κόσμου και έτσι να έχουμε μια παρουσία και σε αυτό το μέτωπο τώρα για το 5G, την πέμπτη, πέμπτη γενιά αυτή είπατε θα κινηθείτε και προς αυτή την ε, κατεύθυνση οπότε να τονίσουμε ότι δεν θα αρκέσουν τα χρηματοοικονομικά μέσα που υπάρχουν για να έχουμε ανταγωνιστικότητα. Ε, το Digital Europe θα απαιτήσει και άλλα μέσα και εργαλεία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλέγμα αποδοτικό κίνητρα φορολογία κατάλληλη οπότε εκτός από τα χρηματοοικονομικά θα πρέπει να δούμε από πάσα από ποιος πώς θα μπορέσουμε να κοντράρουμε με τους παγκόσμιους κολοσσούς. Ο κύριος Μπρετό. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως το καταλάβατε, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, οικοσύστημα, όπως σας το περιέγραψα. Για τα βιομηχανικά δεδομένα να οδηγηθούμε σε παραγωγικότητα όσον αφορά αυτές τις καινούργιες υπηρεσίες το θέμα είναι ποιος θα τα κάνει και ποιος θα ωφεληθεί σήμερα σας είπα γεωπολιτικά τι ισχύει για αυτά τα δεδομένα σε Ανατολή και Δύση που όλοι θα ελκυστούν εδώ θα έρθουν γιατί εδώ θα προσφέρονται όλα αυτά Γι' αυτό και επήγει το θέμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σύμφωνα με το τι ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε κατά αυτό το επόμενο εξάμεινο. Ε, για αυτό και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το οικοσύστημα. Όπως είπατε, να δούμε τι θα κάνουμε με τους ε, γίγαντες, με τις πλατφόρμες, τα προσωπικά δεδομένα ανατομέα, με τους αλγορίθμους. Γιατί μιλούμε και για κάποιους αλγορίθμους που ελέγχουν τα μόρια Οπότε εμείς θα πρέπει έτσι να αναβαθμιστούμε βιομηχανικά και για την αλυσίδα ε, αξίας. Όμως για να μπορέσουμε να γίνουμε γίγαντας θέλουμε την υποδομή ευθύ αμέσω να κινηθούμε από πλευράς δημοσίου κρατικού τομέα για να μπορέσουμε να έχουμε τα μέσα που θέλουμε και να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να οδηγηθούμε και σε αυτούς τους αλγοριθμούς που σας είπα. Άρα είναι ένα πλαίσιο, μια δυναμική για να μπορέσει να γίνει, παραμείνει κυρίαρχη στη βιομηχανία η Ευρώπη. Επομένως εδώ είναι ένα πεδίο μάχης όσον αφορά την βιομηχανία. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Ζωρόν, άκουσα που είπατε τα βασικά προβλήματα όσον αφορά την ψηφική τεχνολογία και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, αλλά έχει αναποφασιστικότητα γιατί δεν ανέλαβε δράση κατά αυτών των γιγάντων του ε, διαδικτύου όσον αφορά τα φορολογικά. Ανελήφθη πρωτοβουλία και 3% ε, πρότεινε η, η Γαλλία για αυτούς τους γίγαντες γιατί κερδίζουν πολύ περισσότερα αυτές οι εταιρείε από όλε τι άλλε στη Γαλλία. Μα πώς είναι δυνατόν αν έχουμε τέτοιο θέμα τον αγωνισμό να τα καταφέρουμε. Οπότε δεν μας εκπλήσει ότι δεν έχουμε προθελτή Ευρωπαίο όσον αφορά τα ψηφιακά και για το 3% είπε ότι ο Τραμπ ε, θα φορολογήσει ε, με 2,4 δις τις γαλλικές εξαγωγές τυρί και κρασί. Μεγάλη ήταν αυτή για την Ευρώπη. Αν επομένω τον όσα δεν κλειστεί κάποια συμφωνία θα βγούμε χαμένοι. Οπότε η Ιρλανδία, Σουηδία και Δανία δεν βοήθησαν τόσο ώστε να τα συμφωνήσουμε και μια που υπάρχει τέτοια εσωτερική αντιπολίτευση, θεωρείτε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που θέλετε να κάνετε. Πώς θα τα κάνετε επίσης, μα πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε αντίπεινα εάν πρόκειται να αυξήσουν οι Αμερικανοί τους δασμούς όσον αφορά τα γαλλικά και τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ κυρία Ζωγόν για την ερώτησή σας. Είναι σαφέστατα τα πράγματα. Σήμερα συζητούμε σε επίπεδο σα για την πρόταση αυτή ε, φορολόγηση σε 154 χρόνια, ε, κράτη. Συγγνώμη. Χαίρομαι που έχουν ε, προχωρήσει πολύ θετικά οι διαπραγματεύσεις. Έχουν συμφωνήσει σχεδόν όλοι, σίγουρα οι ευρωπαϊκές χώρες όλες, αλλά έχετε δει και το υπενήσεστε στην ερώτησή σας, οι Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα δεν έχουν ε, ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία που ελπίζω να γίνει στα πλαίσια του ΩΣΑ. Νομίζω ότι είναι καλή η συμφωνία αυτή που συζητείτε, αλλά φυσικά δεν μπορεί παρά να είναι... Ε, δεν μπορεί να είναι εθελοντική όπως κάτι τέτοιο είχαν προτείνει κάποτε οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, θα πρέπει να είναι ε, δεσμευτικού χαρακτήρα, υποχρεωτικής καταβολής από κάθε φόρος. Ε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία στους όσα ε, συμφωνούν τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης να αγωνιστούν σε περίπτωση που δεν καταστεί αυτό δυνατό, θα την υιοθετήσουμε εμείς και θα την εφαρμόσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να τη διευρύνουμε και εκτός των συνόρων μας. Εγώ είμαι αισιόδοξο για τις συζητήσεις που γίνονται και όπως κατανοούν όλοι και αισθάνονται υπάρχει μια δυναμική. Αναφερθήκατε σε μία από τις χώρες που κατά τα άλλα μου είναι ιδιαίτερα αγαπημένη. Έχει αφήσει κάποιο χρόνο για να καταβάλει ε, το φόρο, μάλλον τον εισπράξει το τελευταίο τρίμηνο, γιατί αυτό είναι και ο χρονικός ορίζοντας των ΩΣΑ. Ο κύριο Κολάγια από τους Πρασίνους ε, στην ΙΜΚΟ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που ήρθατε στην ακρόασή μας ε, μια πολύ, πολύ άσχολη ημέρα όταν βγάλατε αυτές τις τρεις ε, στρατηγικές ανακοινώσεις και ειδικά όσον αφορά την Λευκή Βίβλο για την ε, τεχνητή νοημοσύνη η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των δεδομένων που θα πρέπει να σέβονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτικότητα πρέπει να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπει πολύ θετικά η ομάδα μας και θα ήθελα άρα να σας ρωτήσω αν θα σκεφτόσασταν τεχνολογία η οποία θα μετρίαζε το περιεχόμενο για να αποφευχθούν παραδείγματο χάρη προκαταλήψεις για το φίλο, τη φιλή οτιδήποτε θα μπορούσε να περιλαμβάνει διακριτική μεταχείριση όταν επίσης ε, μιλήσατε στην ακροασή σας για την ψηφιακή στρατηγική είχατε δεσμευτεί για το ότι δεν θα αμφισβητήσετε το καθεστώς μειωμένης ευθύνης των πλατφορμών. Τώρα όμως με το έγγραφο λέτε πως πρέπει να ενισχυθεί η ευθύνη των πλατφορμών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω Εάν μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις για να αποφευχθεί η υπερβολική αφαίρεση περιεχομένου. Απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε ε, ε, Κολαγιά για την ερώτησή σας και σας. Λοιπόν, συγκρατώ δύο σημαντικά στοιχεία από όσα είπατε. Πρώτα από όλα, η παρακολούθηση, ο έλεγχος ε, κάποιου, κάποιου περιεχομένων από κάποιες πλατφόρμες. Οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί για συγκεκριμένες κατηγορίες. Τις γνωρίζετε όλοι, έχετε εργαστεί πολύ από αυτόν. Περιεχόμενο μίσους, υποδάβληση της τρομοκρατίας, ε, παιδικά, παιδική πορνογραφία, fake news, ε, όλα αυτά είναι αρκετά καλά νομοθετημένα και υπάρχουν και υποχρεώσεις. Κατά τα άλλα, πώς να το πω, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι κάποιες πλατφόρμες ε, αρχίζουν και εισάγουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν με τρόπο πάρα πολύ λεπτό να ελέγξουν αυτές τις κατηγορίες, όχι τα πάντα, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουμε πει ότι ε, είναι παράνομη η διάδοση τέτοιου περιεχομένου. Είναι μια στρατηγική προς το παρόν μη ε, δεσμευτική. Θα δούμε πώς θα πάει η εφαρμογή και ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων. Πριν από δύο-τρία χρόνια δεν το είχαμε διανοηθεί καν. Ε, αποδίδουν αυτά 80%, 90% για συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μιλάμε για συνολικό έλεγχο του περιεχομένου. Να είναι σαφή τα πράγματα, σας το είχα πει και το ξαναλέω. Αλλά να έχουμε κάποια μέτρα πλαισίωσης, βοήθειας, ε, ίσως λίγο πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν. Για τις πλατφόρμες μπορούμε να δώσουμε κάποιες υποχρεώσεις συστηματικού χαρακτήρα, χωρίς να αμφισβητήσουμε την ε, εξαίρεση της γενικής ευθύνης από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτησή σας. Γι' αυτό ανοίγει η διαβούλευση και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θα ξανανοίξω την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί και τι δεν μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές ε, εξελίξεις και αυτές που είπατε ίσως και άλλες και πώς δεσμεύονται αυτοί οι μεγάλοι πάροχοι για κάτι που είναι πραγματική υποχρέωση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ευρία απέτηση των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Νίνιστο από τους Πρασίνους συντονιστή στην Ήτρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Πολλά υποσχόμενα αυτά που μας είπατε, ε, αυτές οι προτάσεις της Επιτροπής. Έχετε αυτή την προσέγγιση βάσει των ε, κινδύνων και έτσι να αποκτήσει πρωτοπορία για τα δεδομένα η Ευρώπη, οπότε μπράβο σας. Τώρα εγώ όμως θέλω να τονίσω κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη για τα ψηφιακά. Απουσίασε σήμερα από την συζήτηση η σχέση μεταξύ των ψηφιακών και της νέας πράσινης συμφωνίας. Σημαντικό αυτό από δύο πλευρές. Τι θα γίνει με τα δεδομένα, πώς θα συλλέγονται, με τι τεχνολογίες θα γίνουν όλα αυτά, θα έχουμε ενεργειακή αποτελεσματικότητα, πώς θα περιορίσουμε τις βλαπτικές εκπομπές, πώς θα είναι το ενεργειακό πιο βιώσιμο για να μπορέσουμε να έχουμε και απασχόληση και τεχνολογική πρωτοπορία ε, και λοιπά. Οπότε πάνω σε αυτό θέλω να μας πείτε περισσότερα. Βιομηχάνη δεδομένα για την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα έχουμε κάποιο είδους πρωτυποποίηση των δεδομένων και διαλειτουργικότητας της λύσης έλεγχο της ζήτησης της ενέργειας και άρα να έχουμε και περιορισμό των βλάπτικων εκπομπών. Το 1,4 των εκπομπών έρχεται από τα ψηφιακά σύμφωνα με το Παγκόσμιο Φόρουμ και 7% του ε, ηλεκτρικής ενέργειας και αυτά θα έχουν διπλασιαστεί μέχρι το 2020. θα πρέπει να περιοριστούν οι βλαπτικές εκπομπές με αυτά τα κέντρα διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων με ανακύκλωση και με πρώτες ε, ύλες που θα είναι κατάλληλες για την ψηφιακή τεχνολογία. Σε όλα αυτά ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Πώς λοιπόν θα πορευτούν θα πορευτούν προς αυτούς τους δύο στόχους ψηφιακά δηλαδή και νέα πράσινη συμφωνία σας ευχαριστώ, λέει ο Επιτρόπος. Είναι πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις σας. Πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Αυτά τα δεδομένα και την άλλη μεριά το θέμα του ενεργειακού. Α, πάμε σε ένα εστιατόριο, σε φασφουντάδικο και βλέπουμε όταν υπάρχει διαφορά ε, του μενού Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται όταν πάνε τα παιδιά σας λοιπόν εκεί πέρα για να φάνε ό,τι γίνεται εκεί καταναλώνει πολύ ενέργεια. Οπότε θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Και εμείς τι προτείνουμε. Όσον αφορά τις πλατφόρμες είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση κάθε 18 μήνες αλλά Έχουμε τους μικροεπεξεργαστές και θα πρέπει το ίδιο να γίνει παντού. Και για την επεξεργασία και για την αποθηκεύση των δεδομένων. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνει αυτό η βιομηχανία και υπάρχει βούληση προς τούτο. Να έχουμε τα μέσα και τα οικονομικά και με το Green Deal. Έχετε δίκιο οι βλαπτικές εκπομπές προέρχονται περισσότερο από τα δεδομένα από ότι από τις αερομεταφορές. Άρα, χωρίς τεχνολογία δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε Green Deal. Ούτε να έχουμε τεχνολογία για τα δεδομένα χωρίς το Green Deal. Επομένως, αυτά πάνε χέρι-χέρι. Και κάθε πρόταση που κάνουμε για τις πλατφόρμες θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις επενδύσεις κοινοτικές, κρατικές που θα πρέπει να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που εσείς προδιαγράψατε αλλιώς τίποτα. Κρασνοντέμψκι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε πως ε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα ε, σχεδόν πάντα προσπαθούν ε, να μειώσουν τις διαφορές ε, μεταξύ των ε, κυβερνήσεων. Γιατί Βεβαίω είναι διαφορετικές εξελίξεις χωρίς την συνέργεια. Θεωρώ λοιπόν πως τα νέα προγράμματα στον δικό σας τον τομέα, τεχνητή νοημοσύνη και τα σχετικά, θα πρέπει να περιέχουν το στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν ερευνητικά έργα στον διασυνοριακό τομέα. Πρέπει να διασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία για να μην διαταραχτεί η πολιτική των επενδύσεων. Μία περσινή έκθεση της McKinsey δείχνει πως ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ετοιμότητα για τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ε, θέλει να αντιμετωπίσει λοιπόν η Κομισιόν το πρόβλημα αυτό. Έχετε προγραμματίσει κάποιους μηχανισμούς συνοχής ή όχι. Θεωρώ πως ε, εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος ε, τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Ο κίνδυνος δηλαδή λόγω της ψηφιακής επανάστασης να έχουμε ξανά έναν διχασμό της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Κρασνοντέψκη για την ερώτησή σας. Για την απάντηση ανοίγετε κι εσείς μια προοπτική εδώ. Θα πάω να συνεργαθώ με τη συνάδελφο που ασχολείται με τα θέματα συνοχής. Πολύ καλή ιδέα για τον προπολογισμό. Θα την αδράξω αμέσως. Ε, ακόμα και αν το σχέδιο που εμείς ε, προτείνουμε είναι ένα σχέδιο το οποίο εξορισμού είναι διασυνοριακό, cross border στα αγγλικά. Αφορά όλες τις αλυσίδες παραγωγής αξίας ε, και αγκαλιάζει όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είπα ότι αρχίζαμε ε, από ότι μας επέτρεπε να έχουμε αυτή την ε, ισχύ υπολογιστών ε, με το HPC, τον, τον υπερυπολογιστή τον ευρωπαϊκό και το ανοίγουμε σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχει ήδη αυτή η υποδομή, δεν ε, είναι αποκλειστικότητα ενό ή δύο κρατών. Όποιο θέλει από εκεί έχει πρόσβαση. Γι' αυτό σα είπα ότι θα χτίσουμε αυτά τα τουβλάκια για να μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν χωρί ε, να παραμείνει κανεί πίσω. Να αφορά όλα τα κρατημέλη, όλους τους κλάδους για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και το δεύτερο στοιχείο, σας το είπα και το ξαναλέω, στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε δομές πλαισίωσης ε, ανακλάδου παραγωγής, αναλυσίδα παραγωγής αξίας. Όπως σας είπα, ε, ε, ε, κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες θα επωφεληθούν σε τοπικό επίπεδο με συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη σε εκείνους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια όπου και να βρίσκονται στην Ευρώπη. Θα τους βοηθήσουμε για να μπορέσουν καλύτερα να αξιοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία και να χρησιμοποιούν είτε τα δεδομένα που θα παράγουν οι ίδιοι, είτε κάποιους αλγόριθμους που κάποιοι άλλοι θα έχουν ε, δημιουργήσει και θα τους ε, παρέχουν. Αυτό το πουλ, το σύνολο των δεδομένων που είναι δημόσια, ανώνυμα, θα στρέφεται κατά κύριο λόγο και κατά προτεραιότητα σε όλες τις μικρομεσαίες και τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κυρία Μπέτα, Μπεάτα Μαζούρεκ, ε, ε, ECR IMCO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, εσείς ε, και οι συνεργάτες σας στην Κομισιόν είπατε πάρα πολλά πράγματα για την αναγκαιότητα της ψηφιακής επανάστασης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είπατε πως θα πρέπει οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείε να παίξουν ένα ρόλο κλειδί και επιπλέον γνωρίζουμε πως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από εταιρείε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς ε, την στήριξη αυτή δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Το νέο πρόγραμμα δείχνει πως η Κομισιόν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα όμως ε, να αναφερθώ στα διάφορα έργα που υπάρχουν και έχουν ήδη αποτελέσματα. Τέτοια έργα υποστηρίζουν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα σχέδια στον ε, τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Μιλάμε για ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα, καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ, στήριξη της Τελωνιακής Ένωσης και πράσινο deal. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, το GovTech λέγεται, το οποίο αφορά τις δημόσιες προμήθειες, υποστηρίζει την ψηφιοποίηση. Ε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία, Πολωνία και αλλού και προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία η οποία ακόμα δεν έχει εξαντληθεί. Δεν την χρησιμοποιούμε πλήρως. Λοιπόν, μπορούν να είναι καινοτόμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η GovTech. Θα δώσετε κάποια ευκαιρία λοιπόν στις ε, εταιρείες αυτές να γίνουν οι πρωταθλητές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Είναι τεράστιο το πεδίο αυτό και η ερώτηση που ε, μου θέσατε κυρία Μαζούρεκ. Επανάσταση είναι, δεν ξέρω, εξέλιξη είναι. Δεν μου αρέσει ο όρος revolution, χρησιμοποιώ το, όρο evolution. Είναι μια εξέλιξη, όπως και η Πράσινη Συμφωνία, ε, θα εξελιχθεί, θα ξεδιπλωθεί μέσα στην επόμενη 25 ετία. Υπάρχει ο, ο ανθρώπινος χρόνος, η εκμάθηση, είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, θα χρειαστεί χρόνο, δεν θα γίνει σε μια διετία. Τις αποφάσεις όμως τώρα πρέπει να τις πάρουμε, αυτό είναι σίγουρο. Και με κάποιες εφαρμογές που μπορεί να έχουν σημαντικές ε, επιπτώσεις. Ε, επαναλαμβάνω, για τα δημόσια δεδομένα θα φροντίσουμε να έχουν πρόσβαση ε, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες και άλλα δεδομένα για τις δημόσιες υπηρεσίες επίσης βελτιώνεται. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω δει πολλούς υπουργού από κράτη-μέλη που μου έλεγαν ότι «Α, τώρα θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο εργαλείο για να συλλέγουμε καλύτερα τους φόρους. Αυτό το έχω ζήσει εγώ στο πετσί μου, γιατί έχω διατελέσει υπουργό Οικονομικών. Σε όλες τις χώρες υπάρχει φόρο διαφυγή, που θα πρέπει να πατάξουμε για να αυξήσουμε τα οικονομικά μας έσοδα, τα φορολογικά έσοδα που τα έχουμε και ανάγκη. Και εδώ χρειάζονται φυσικά ε, άνθρωποι προσωπικό, αλλά και αλγόριθμοι πιο περίπλοκοι για να μπορούμε να εντοπίζουμε τους φοροφυγάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούν λοιπόν οι δημόσιες διοικήσεις τώρα να είναι πιο αποδοτικές, πιο αποτελεσματικές. Ε, αυτό φυσικά δεν καλύπτεται ε, από τη στενή έννοια από τη σημερινή μου παρουσίαση, αλλά το υπενήσετε αυτό, γιατί κάθε οργανισμός που παράγει δεδομένα μπορεί να τα χρησιμοποιεί στη συνέχεια για να εξυγχρονίζεται, για να βελτιώνεται και να είναι και καλύτερο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να καινοτομεί κτλ. Και φυσικά στις δημόσιες υπηρεσίες τελικά θα παρέχουν καλύτερη υπηρεσία σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουντούρα, παρακαλώ, από την ΚΟΕ ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπρετόν, σχεδιάσατε να ρυθμίσετε την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ακολουθώντας ένα μοντέλο που βασίζεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητάς της Ωστόσο, οι εκτιμήσεις κινδύνου που επικαλείστε, παρόλο που είναι πολύτιμες, δεν μπορούν να αξιολογήσουν σημαντικές απειλές στην αυτονομία, ελευθερία, ιδιωτικότητα και άλλες βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα του ατόμου, καθώς για αυτούς τους κινδύνους δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα οι κατάλληλες μεθοδολογίες. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό κατά την εφαρμογή του πακέτου που μας αναφέρατε. Έχουν επίση εκφραστεί σοβαρέ ανησυχίε για του κινδύνου που ενέχει η χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα των τεχνολογιών αναγνώριση προσώπων σε δημόσιου χώρου. Εγώ θέλω να προσθέσω την ανησυχία μου για τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη στου χώρου εργασία, δεδομένου ότι η φυσική παρακολούθηση τη φυσική συμπεριφορά και τη αποδοτικότητα των εργαζομένων και η αθέμητη επεξεργασία δεδομένων στην εργασία την καθιστά αδικαιολόγητη και παρεμβατική τι προτίθεστε να κάνετε για να ρυθμίσετε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των προσωπικών τους δεδομένων. σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού η Ευρώπη δέχτηκε 577 εκατομμύρια επισκέψεις το 2019, οι οποίες έφεραν πάνω από 400 δις ευρώ εισόδημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική δύναμη και επίσης είναι ο μεγαλύτερος επιταχυντής ανάπτυξης θέσεων εργασίας παγκοσμίω. Γνωρίζω ότι έχετε προτεραιότητα τον τουρισμό και αναφέρατε μάλιστα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν σχεδιάζει η Επιτροπή να ενσωματώσει τον κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία τομέα του τουρισμού στην ιεράρχηση των πόρων για την έρευνα τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων γιατί εκτός από απολύτως απαραίτητο είναι και κοινωνικά αναγκαίο. Thank you very much. Je vous Monsieur Ευχαριστώ. Κυρία Κουντουρά. Ναι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς. Αυτές είναι οι αξίες που θέλουμε και να είναι σύμβατοι η σχετική και όσον αφορά τη συμπεριφορά ή την ατομική συμπεριφορά. Ακριβώς έτσι. Σε αυτό το μέτωπο θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς όπως προανέφερα. Τέτοιου είδους εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση οι αξίες των αλγορίθμων να είναι με τις αξίες μας σύμβατες. Όπως ξέρετε υπάρχουν περιπτώσεις για την οργάνωση, για την αναγνώριση, για τα αεροδρόμια, υπάρχουν προβλέψεις και καλύπτονται από την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος, ένα μορατόριο για να δούμε πώς αυτή η αναγνώριση ναι, χρειάζεται προσπάθεια φυσικά και δεν επιτρέπεται γενικά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε ε, κάποιο δωμάτιο με ασφάλεια ε, για νοσοκομεία κλπ. Ήδη υπάρχει όμως νομοθετική πρόβλεψη. Αποδίδει. Και να δούμε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνολογία. Τον τουρισμό βεβαίως και έχει μεγάλη δυναμική. Είναι σημαντικός ο κλάδος αυτός. Σαφώς είναι σπουδαίο θέμα και εκεί είναι μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας ο τουρισμός. Έχουμε τώρα νέες αρχές και εκεί έχουμε αλγορίθμους και για να είμαστε ξεκάθαροι όχι, εκεί δεν θα υπάρξει ε, καθυστέρηση. Βεβαίως θέλουμε ένα περιθώριο για να το ψάξουμε αλλά θα πρέπει να γίνει προσαρμογή. Η κυρία Σοφή Πελτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Η στρατηγική σας έχει φιλοδοξία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στα ψηφιακά εργαλεία, τα σημερινά και τα μελλοντικά. Έλεγε ο Κορνέη ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη ε, προσελκύει τον κίνδυνο. Και είναι μεγάλη καχυποψία και σωστά ο κόσμος φυλάσσεται. Η ε, εμπιστοσύνη κατακτάται, αλλά δεν αποκλείει τον έλεγχο. Θα πρέπει οι πλατφόρμες να σέβονται το δίκαιο, να πληρώνουν τους φόρους τους, ανάλογα με τα κέρδη, να μην υποφελούνται από τη δεσπόζουσα θέση. Δεν είναι η λογική εδώ ο ανταγωνισμός, αλλά οι αξίες η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η διαφάνεια, η δεντολογία θα πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών και εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και λογική. Πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε την προστασία των δεδομένων, γιατί τα δεδομένα, τα data τώρα τα λέτε σαν να είναι το καινούργιο Αλντοράδο. Στην υγεία που γνωρίζω καλά, ε, τα ιατρικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο νέο μαύρο χρυσό ε, τα ιατρική λήψη ψηφιοποιημένη θα πρέπει να είναι ε, προστατευμένη και να είναι ιερό το θέμα της προστασίας ε, των προσωπικών στοιχείων. Σε όσα είπε η κυρία Κουντουρά για την αναγνώριση προσώπου, χρησιμοποιείται ήδη και ο κόσμος ανησυχεί. συμφωνούμε όλοι ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η ψηφιακή αυτή μετάβαση και στη σας θεώρηση ε, δεν καταλαβαίνετε τι ε, γίνεται ε, και πώς είναι οι εργασιακές σχέσεις στον Deliveroo, στο Uber, στην Amazon. Είναι νέα σκλαβιά πλέον, δεν είναι εργασία αυτή. Και σας ερωτούμε, ποιο είναι το τίμημα όλων αυτών, οι ελευθερίες, τα δικαιώματα, η αρχή της προφύλαξης, της ισότητας, συστηματική παρακολούθηση, καταστολή οι Ευρωπαίοι χρειάζονται, ε, κύριε Επίτροπε, συγκεκριμένες και διαφανείς εγγύησεις. Απάντηση. Ευχαριστώ, κύριε Πελτσιέ. Ακούγοντάς σας, και μην με παρεξηγήσετε την αρχική σας τοποθέτηση, αναρωτήθηκα, δεν ήσασταν ε, δίπλα μου όταν συναντήθηκα με τον πρόεδρο ε, μήπως είσαστε δίπλα μου μάλλον όταν συναντήθηκα ε, πρόσφατα με ένα πρόεδρο μιας μεγάλης ε, ψηφιακής εταιρείας. Ακριβώς τα ίδια του είπα, επιλέξει. Ε, φυσικά αυτά με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και όσοι έρχονται να μας δουν, αυτά ακούν, αυτά τους λέω για τις πλατφόρμες, για τη δεσπόζουσα θέση, για τον αντίκτυπο στην αγορά, για τις ευθύνες τους, για την κοινωνική τους ευθύνη. Μάλιστα τους είπα νομίζω ότι οτιδήποτε δεν απαγορεύεται, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται αυτομάτως στο σημερινό μας κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο. Ε, υπάρχουν κοινωνικές ευθύνες που θα πρέπει να μοιραζόμαστε. Και φυσικά, ε, συμφωνώ απολύτως και γράφαμε στο πλαίσιο των όσων είπατε. Ε, εκεί θα εργαστούμε τους επόμενους μήνες και στην Ομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα σας καταθέσουμε στα τέλη του έτους την πρόταση. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα τον όρο μαύρος χρυσός. Δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος, γιατί τα δεδομένα είναι γεγονός. Είναι δεδομένο, για να το πω έτσι. Εμείς θα πρέπει να οργανωθούμε στην υγεία. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να προστατεύονται απολύτω ε, με ανώνυμο τρόπο, ε, τα στοιχεία των ασθενών, φυσικά με πάρα πολύ ακριβή και προσεκτικό τρόπο και πάντα ε, εθελοντικά. Επίσης, συμφωνώ για τα δεδομένα υγείας, σας είπατε. Και κατά τα άλλα αυτό ισχύει και όταν θα χρησιμοποιούμε αλγορίθμους που μπορούν να μεταφερθούν εκτός της Ένωσης και για αυτά τα κρίσιμα στοιχεία της υγείας. Εγώ όμως ήμουν εκείνος που σας είπα μαζί με κάποιους συναδέλφους της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία που παίρνουν οι αλγόριθμοι μαζί τους εκτός της Ένωσης και στην υγεία. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα πράγματα να ξέρουμε ποιο είναι πίσω από τον αλγόριθμο. Υπάρχουν κρίσιμε εφαρμογέ που πρέπει οπωσδήποτε να τι προσέξουμε. Αναφερθήκατε σε μια μορφή σύγχρονη δουλεία. Σα είπα στην εισαγωγή μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των εργασιακών συνθηκών και το εντάσσουμε απολύτω στην πολιτική μα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε δέκα ομιλητές ένα λεπτό καθένας και στο τέλος θα ζητήσω από τον κύριο Επίτροπο να απαντήσει σύντομα εντός πέντε λεπτών. Ξεκινάμε την κυρία Εύα Μαϊντέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Ε, καμιά φορά χαίρεται κανείς που είναι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως σήμερα. Γιατί τα τρία έγγραφα τα οποία παρουσιάσατε ε, δεν αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα σημερινό ή χτεσινό ή αυριανό. Αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολεί για κάποια χρόνια, αλλά κάτι το οποίο είναι σημαντικότερο, είναι ένα θέμα του μέλλοντος που θα μας απασχολεί στα επόμενα 10-20 χρόνια και παραπέρα. Ένα ζήτημα ε, το οποίο θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις οικονομίες μας, ε, θα μας δώσει καθαρή τεχνολογία. Εγώ το θεωρώ ε, ένα είδος ρύθμισης που θα βοηθήσει την εφευρετικότητα. Χαίρομαι λοιπόν ότι δώσατε ιδιαίτερο βάρος στα δεδομένα. Μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά τον διαμοιρασμό δεδομένων. Προβλέπετε νομοθεσία μέχρι το τέλος του έτους. Δώστε μας λίγες περισσότερες λεπτομέρειες και καταλήγω για να είναι πλήρη αυτά τα έγγραφα πρέπει να εκφραστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να πείστε τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ κυρία Κοταγιάρ. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Η Ευρώπη έχει ένα μοναδικό μοντέλο κοινωνικής οικονομίας αγοράς το οποίο μας κάνει υπερήφανους και επέτρεψε στην Ένωσή μας να αναπτυχθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη, ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και δικαιώματα των πολιτών. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να επικαιροποιήσουμε αυτό το μοντέλο και να πάμε προς μια ψηφιακή κοινωνική οικονομία της αγοράς. Πριν από λίγες ε, μέρες ο κύριος Βόλφ, διευθυντής ενός Think Tank ε, ονόματι Μπρούκελ, είπε ότι η Ευρώπη θεωρεί εαυτόν τον διαιτητή του ψηφιακού κόσμου, αλλά οι διαιτητέ δεν κερδίζουν. Και εγώ θα προσέθω ότι μόνο το βρεσίδι ακούν. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τους κανόνες και μετά να παίξουμε και το παιχνίδι. Όσον αφορά λοιπόν την ε, τεχνητή νοημοσύνη, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Αλλά ως γενική παρατήρηση θα έλεγα ότι η πολιτική μας οικογένεια θα είναι ιδιαίτερος ε, προσεκτική όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Πρέπει να δούμε την δεοντολογία και τα δικαιώματα φίλου ατόμων με αναπηρία και ευπαθών ομάθων. Σας ευχαριστώ κύριε Μπότος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην ε, συνεδρίαση των επιτροπών μας. Μιλήσατε για το ότι θα προσπαθήσετε να βελτιώσετε τις πτυχές ε, του εμπορίου. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει διάφορους ε, κανονισμούς. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό ε, να είναι κάποιος υπεύθυνο για την ασφάλεια των προϊόντων και τα σχετικά. Αλλά στην ψηφιακή αγορά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Το είπατε κι εσείς. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ο καταναλωτής. Δεν υπάρχει ένας υπεύθυνο για την συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών για προϊόντα που αγοράζονται στο διαδίκτυο και κατασκευάζονται σε τρίτη χώρα. Το πρωτόκολλο λοιπόν που έχει υπογράψει με τι πλατφόρμες δείχνει καλή βούληση και από τι δύο πλευρές, αλλά πρέπει να ρυθμιστεί ο κλάδος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η πρωτοβουλία για την ψηφιακή αγορά θα περιλαμβάνει έναν σαφή μηχανισμό που θα καθορίσει την ευθύνη και την αστική ευθύνη των ε, πλατφορμών. Και πότε νομίζετε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιο μηχανισμό. Ο πρόεδρος, σας παρακαλώ ε, να τηρείτε το χρόνο, έχουμε 20 συναδέλφους. Κύριος Παύλο Αρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, όσον αφορά τον αθλητισμό, αυτός που είναι προπονημένος ξεκινάει πρώτος έχει πλεονέκτημα και αυτός που παίρνει την τόπα. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει όσον αφορά την διαφάνεια. Έχει τέτοιο πλεονέκτημα όπως ο αθλητής που το πάρετε. Για μας όμως ε, αυτά που κάνει η Αμερική είναι κόκκινη γραμμή. Άρα θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και επομένως θα πρέπει να είμαστε ευφυείς και καινοτόμοι. Θα πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμε λύσεις, οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια οι ΜΜΕ που έχουν εμπειρία και την τεχνολογική γνώση. Από τις αρχές μας και τις αξίες μας θα πρέπει να δουλέψουμε και να έχει ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη, να έχει διαφάνεια και σεβασμό στον ιδιωτικό βίο. Ε, ο κύριος Ζων Λα Λακαπέλ. Δεν είναι εδώ. Και πάμε στην Κιμ Φαν Σπάρεντακ. Είναι εδώ ο κύριος Λακαπέλα. Ε, ε, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Συμφωνούμε ε, για το ρυθμιστικό πλαίσιο, για τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου. Ε, εκτός αυτού όμως θα υπάρξει και εθελοντική ρύθμιση για τις ε, εφαρμογές μη υψηλού κινδύνου. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία τώρα. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Αν ανημερωθεί, αν ανανεωθεί, δεν μπορεί να καλύπτει την προστασία των καταναλωτών. Ή ε, καλύπτει ε, ακριβώς την προστασία, τότε δεν χρειάζεται εθελοντική ρύθμιση. Ε, ο χαμηλός κίνδυνος δεν σημαίνει μηδενικός κίνδυνος, ας πούμε στα παιχνίδια για βρέφη. Ε, γιατί να είναι διαφορετικό για την τεχνητή νοημοσύνη αυτό που ακολουθούμε. Ευχαριστώ. Επανα... Επανέρχομαι στον κύριο Λακαπέλ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που επιβεβαιώνει ότι ψηφιακός κλάδος στην Ευρώπη υπό αναπτύσσεται. Η Ευρώπη αδρανεί και η Αμερική ε, επελάβνει στις αγορές μας. Γκάφα, Google, Amazon, Facebook, Apple είναι αποκλειστικά αμερικανικές εταιρείες. Τώρα ε, έρχονται οι Κινέζοι που προσπαθούν να βάλουν εδώ την τεχνολογία 5G με τεράστιους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια. Ανισχυτικές εξελίξεις και τεράστιο το πρόβλημα ε, για τις εξωτερικές επιχειρήσεις ξένες που κυριαρχούν εδώ και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν τις καθορίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμώνεται για ποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε τους δικούς μας ε, πρωταγωνιστές στη ψηφιακή οικονομία. Θυμίζω ότι το 70 η Airbus ε, δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί την Boeing και σήμερα είναι ο επαριθμόν ένα κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο και είναι ευρωπαϊκός ε, πρωταθλητής. Θα χρειαζόμαστε μια δική μας Silicon Valley στην Ευρώπη έτσι ώστε οι μικρομεσαίες και οι να ευημερούν. Χρειαζόμαστε τη μεγάλη Ευρώπη της βιομηχανικής συνεργασίας αυτή που μας επέτρεψε να ε, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στην αεροναυπηγητική. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που θα πάρετε και πώς θα έχουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές ε, στα ψηφιακά. Η κυρία Λετάου Μάρκες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι ευχαριστώ τώρα σήμερα σε σχέση με αυτά τα οποία διαβάσαμε στα έγγραφά σας για η στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε πώς θα αναπτυχθεί ούτως ώστε να βελτιωθούν οι κρατικές υπηρεσίες και από εκεί έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε να κερδίσουμε τελικά για την ψηφιακή αλλαγή την εμπιστοσύνη του κόσμου και σας ερωτώ είναι δυνατόν αυτά τα δεδομένα να τα σωρεύσουμε, να τα φιλτράρουμε από τον ιδιωτικό τομέα. Με τι στρατηγική θα το κάνετε αυτό. Πώς θα μπορέσει το δημόσιο να αντιλήσει, να αξιοποιήσει τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα. Ε, αν θέλετε μπορείτε να μου απαντήσετε αργότερα. Ε, χρειάζεται όμως και κάποια συνενετική στρατηγική για τις ε, ιντερνετικές πλατφόρμες αυτές. Είναι ε, μονοπόλια. Τι θα γίνει. Ε, ε, ο επόμενος κυρία Πιλάρ Ντελγαστή, ευχαριστούμε για αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα καθοριστεί έτσι η πολιτική μας την επόμενη πενταετία. Πρώτα-πρώτα είναι ε, πολύ βασική την ετοιμοσύνη, προχωρημένοι υπολογιστές και να υπάρχει μια τέτοια βάση δεδομένων, αλλά χρειάζεται υποδομή. Συγκεκριμένη με ερώτηση. Ήδη στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα έχουμε το νέφος, μπορούμε αυτά να τα συνδυάσουμε, οπότε δεν χρειάζεται να φτιάξουμε ένα άλλο νέφος, να αρχίσουμε από το μηδέν. Αν αυτό ισχύει, τότε θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την διαδικασία αυτή, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο τρίμηνο του 22 και να μην ξεχνούμε και εδώ επικαλούμε αυτά που έχει πει η Κομισιόν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας για το επόμενο ε, διάστημα των πέντε ετών. Η κυρία Τζέσικα Στέγκρουτ. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ που παρουσιάσατε τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σας. Προφανώς είναι ακόμα στο μακροεπίπεδο και όχι στο επίπεδο της ε, νομοθεσίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αυστηρή νομοθεσία προστασίας δεδομένων ε, έχει πολλά μειονεκτήματα για τον κλάδο μας και τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο χωρίς να εγκαταλείψουμε αυτές τις υψηλές προδιαγραφές. Θεωρώ όμως ότι τελικά το θέμα αυτό θα προσθέσει περισσότερες ρυθμίσεις παρά θα στηρίξει την καινοτομία. Οι ψηφιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν άγριο παγκόσμιο ανταγωνισμό και προφανώς η αμερικανική προσέγγιση είναι πάρα πολύ επιτυχής. Από τις 100 κορυφαίες εταιρείες, μόνο 12 έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 45 έχουν έδρα στη ΣΥΠΑ. Πώς μπορείτε να μην πείσετε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος δρόμος, μια που αποφασίσατε να μην αντιγράψετε, ούτε καν να διδαχτείτε από το πιο επιτυχημένο μοντέλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λέει η κυρία Γκαμόν. Χαίρομαι που αναφέρατε την ασφάλεια. Είχατε πάει και σχετική διάσκεψη του Μονάχου. Αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι δεν υπάρχει μια ολιστική ε, αντιμετώπιση της ε, στρατηγικής. Καλοδεχούμε λοιπόν η νέα προσέγγισή σας. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στην ε, Ήτρε είναι το κέντρο για την κυβερνοασφάλεια. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς να ενσωματώσετε την διάσταση της έρευνας. Θεωρείτε ότι το κέντρο αυτό είναι ένα καλό μέτρο και πώς ακριβώς εντάσσεται στην στρατηγική σας. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο βεβαίως να παρακολουθεί κανείς το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις ειδικά σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, έχετε πέντε λεπτάκια, αν μπορείτε. Α, πάρα πολύ ωραία. Πριν μου δώσατε δύο λεπτάκια, τώρα πέντε ολόκληρα. Α, ναι, ναι, σωστά, σωστά ήταν και περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, επανέρχομαι σε κάτι σημαντικό. ακριβώς ε, το πώς θα διαχειριστούμε τον διαμερασμό των δεδομένων. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικά δεδομένα. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχει μια σχετική διαχείριση. Ε, ακριβώς για να υπάρχει μια ε, πιο οριζόντια αντιμετώπιση του διαμοιρασμού, της ανωνυμοποίησης, της επαναξιμοποίησης των δεδομένων. Ε, πρόκειται προφανώς λοιπόν για ε, ένα πλαίσιο οριζόντιο προφανώς ε, και αυτό το οποίο μετά λέμε χώρο δεδομένων και μετά το 2021 θα έχουμε το νομοθέτημα περί δεδομένων για την χρήση από εταιρείες και δημόσιες αρχές. Αυτά προβλέπονται στον νόμο περί δεδομένων. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Το λέω γιατί συχνά τίθεται το ερώτημα. Η κοινωνική διάσταση, η διάσταση της ισότητας του φύλου, όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αντιμετωπίζονται πάρα πολύ εύκολα όταν ξέρουμε τι θέλουμε. Και ξέρουμε άπα και είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να στήσουμε αυτή την αλυσίδα ούτω ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους ε, αλγορίθμους αυτούς που εμπλέκονται στο θέμα και ο ε, καταναλωτής και η προστασία υπάρχει ήδη πλέγμα προστασίας νομοθετικό αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη να τα συγχρονίσουμε και ακριβώς χάρη, χάρη σε αυτούς τους ε, αλγορίθμους Ακόμα υπάρχει να σε ένα παιχνιδάκι ισχύει αυτό. Και στο παιχνίδι επομένω περιέχονται οι αλγόριθμοι, οπότε αυτό μπορεί να επαληθευθεί με την πιστοποίηση. Τα ξέρουμε στη γενική μας ε, διεύθυνση και θα τα προσαρμόσουμε ναι, στο μέτρο του δυνατού τώρα για τη διαφάνεια και τις Ηνωμένε Πολιτείε που εντό σέβονται και την Κίνα. Κοιτάξτε, θα ρυθμίσουμε τις συνέπειες να αξιοποιηθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι γίνανε οι γίγαντες. Αλλά πολλοί θα θέλανε να εκμεταλλευτούν αυτή την ε, πρωτοπόρα ή μονοπωλιακή θέση, αλλά πρόκειται για την βιομηχανία πρόκειται για κάτι διαφορετικό μια επιχείρηση ας πούμε τα, ξέρετε μιλάμε για επιχείρηση 35-40 εργαζομένων πολυευρωπαίοι και μιλάμε για τριψήφιους αριθμούς μηχανικών και ξέρω καλά και τις δύο πλευρές. Αυτοί έχουν το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις. Οπότε έτσι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενοι τα βιομηχανικά δεδομένα να πάνε μπροστά. Πιέζει ο χρόνος. Μίλησε με την πέμπτη γενιά, 5G, κυβερνοασφάλεια, σημαντικό, η ασφάλεια ορίζουν νομοθεσία για την καινοτομία. Όχι, δεν θα κάνουμε ότι οι Αμερικάνοι. Δέκα χρόνια, δέκα δις. Ούτως ώστε αυτοί δεν μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμεί σε σχέση με τις ε, πλατφόρμες. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Εμείς ξέρουμε σήμερα στην ε, Κομισιόν τι γίνεται. Και εσείς να το ξέρετε αυτό ξεκάθαρα. Ποιο είναι το μήνυμα. Είναι το μήνυμα που μπορεί να φαίνεται αισιόδοξο. Άρα θα πρέπει χωρίς αφέλεια να προχωρήσουμε μαζί και να αφουγκραζόμαστε όχι αυτούς που λένε ότι χάσαμε τον πόλεμο. Χάσαμε μία μάχη. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για αυτήν την εκ των υστέρων νομοθεσία. Να έχουμε όσο γίνεται πιο στεγανό πλαίσιο. Συμπαραγωγή. Αυτό θα γίνει τα επόμενα τρία χρόνια. Um, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μπορούμε να συνεχίσουμε ε, λίγο παραπάνω μετά τις 6 και ήδη ευχαριστώ τους διερμηνείς γι' αυτό. Μόνο εάν τηρήσουν όμως αυστηρά το ένα λεπτό που έχουν οι επόμενοι μελητές. Η κυρία Πένκοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κύριε Βρετών για την παρουσίασή σας και για την ψηφιακή ατζέντα. Συμφωνούμε όλοι ε, ε, για τα ωφέλη μάλλον των νέων τεχνολογιών και της οικονομίας των δεδομένων. Θα πρέπει όμως να έχουμε ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Γενική Διεύθυνση Connect και η ε, άλλη Γενική Διεύθυνση που συνεργάζονται πρέπει να ρυθμίσουν κάποια πράγματα. Η φύσμα είναι και ο Επίτροπος Δομπρόφσκης ε, υπάρχουν προτάσεις ή προθέσεις για κοινή νομοθεσία που προτίθεστε να κοινοποιήσετε. Γνωρίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ε, ξεκινάει να ε, αναθεωρεί την οδηγία NIS. Ιδιαίτερα αυτό τι σημαίνει για τις εθνικές αρχές και για τους ε, φορείς ε, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών υπηρεσιών. Κύριε Κλούν, ε, ευχαριστώ που ήρθατε πρόεδρε και για όσα είπατε για τα ανώνυμα στοιχεία υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να το έχουμε υπόψη μας. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικέ πλατφόρμες ευρωπαϊκές για διαμοιρασμό των στοιχείων με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, ιδιαίτερα το θέμα της χρηματοδότησης. Καλό είναι να το εξασφαλίσετε. Ποιε θα είναι αυτές οι πλατφόρμες, πώς θα είναι, ποιος θα τις διαχειρίζεται, πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα και τι θα γίνει με την, ε, την εξαγωγή, ας πούμε, δεδομένων, τον εντοπισμό τους θα πρέπει να είναι μεγάλη η προστασία και των καταναλωτών στα πλαίσια της ε, τεχνητής νοημοσύνης και της νομοθεσίας. Ήδη έχουμε και μεταξύ αυτών είναι και ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αρκούν αυτοί οι νόμοι που έχουμε για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των πολιτών. Η πρόεδρο Φόντερ Λάιν είπαν ότι ε, αν έρθουν νέε νομοθετικέ προτάσει, θα αντικαταστήσουν κάποιε άλλε. Ο κύριο Μπελαμή, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σα. Πολλά έχουν υποθεί ήδη. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο μόνο. Το είπατε και όλοι το υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό. Το αισιόδοξο μήνυμά σα δεν έχει χάσει η Ευρώπη την τεχνολογική μάχη. Ωστόσο οι πολίτε σήμερα θεωρούν ότι άλλοι καθορίζουν το μέλλον και μάλιστα το μέλλον τη Ευρώπη. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να γράψουμε ήδη την ιστορία μας και σε μεγάλο βαθμό την ιστορία της παγκοσμιοποίησης, αντί να την ε, υφιστάμεθα. Για την 5G ιδιαίτερα, η κινητή ε, τεχνολογία 5G δεν είναι 4G με μεγαλύτερη ταχύτητα, είναι νέα αρχιτεκτονική. Εμείς πώς θα μπορούμε να χτίσουμε τους Ευρωπαίους πρωταθλητές, τι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε σήμερα, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πολιτική ανταγωνισμού Πώς θα διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Από τη μια θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί στον ανταγωνισμό για τα καλύτερα προϊόντα για τους καταναλωτές, ταυτόχρονα όμως να έχουμε μια στρατηγική που να εξασφαλίζει την κυριαρχία μας. Δεν θα σας πω ονόματα επιχειρήσεων, όλοι έχουμε υπόψη μας, ε, καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Η, κυρία Στοφαγγλέρη. Μισάριο. Έχουμε τις νέες ε, τεχνολογίες. Μπορούμε να μαζέψουμε όλων τα δεδομένα. Μεγάλη ευκαιρία αλλά και κίνδυνος. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να προβληματιστούμε τι κίνδυνος υπάρχει για τα δεδομένα τα δικά μας εάν ε, εμπιστευτούμε μόνο τα εργαλεία των άλλων να δούμε τι θα γίνει με τις δικές μας επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο, να τις υποστηρίξουμε, τεχνολογίες να γίνουν αυτόνομοι και έτσι η Ευρώπη να μην πέσει στον αυταρχισμό, στο, στο ζυγό των ε, τρίτων. Οπότε θα πρέπει αυτό που λέτε να παίξει σημαντικό ρόλο. Οι ΜΜΕ δυσκολεύονται για να έχουν πρόσβαση ε, στα δάνεια. Άρα τι μπορείτε να κάνετε ούτως ώστε να τις διευκολύνετε να μπορούν να δανειστούν χρήμα για να είναι ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ, Μπουσλάγκα. I recommend really not to call data oil uh, because then... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν οι εταιρείε μας να μοιραστούν τα δεδομένα. Έχω δύο ερωτήσεις από τη σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λοιπόν, εάν σκεφτούμε το τι έκανα εγώ, έφτιαξα μια πολιτική μικρή εταιρεία και ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να τα συμβάσουμε αυτά με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων. Χρειαζόταν δικηγόροι ε, πώς μπορούμε να διδαχτούμε λοιπόν από αυτά έτσι ώστε να μπορούν να συμμορφωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άλλο ερώτημα είναι κάπως πιο προκλητικό. Γιατί επιλέξατε την κυριαρχία ε, αντί για την ανταγωνιστικότητα σε όλα τα έγγραφα. Δηλαδή από τη σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εγώ θέλω μια αριθμισμένη αγορά υπηρεσιών του νέφους, να υπάρχουν αρκετοί παίκτες και να έχω καλές υπηρεσίες, αλλά γιατί πρέπει να φτιάξουμε ε, μια διαφορετική υποδομή από την σκοπιά του κράτους. Σας ευχαριστώ κυρία Μαλτονάλντο Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, σε σχέση με κάτι που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση για τις πλατφόρμες και τη διασύνδεση με την εσωτερική αγορά. Στο σημερινό σας έγγραφο ε, για τα ψηφιακά αναφέρατε ότι Πολλά από τα προϊόντα που εισάγονται στην εσωτερική μας αγορά και είναι πλαστά, είναι παράνομα, ε, ε, απειλούν την ενιαία αγορά που θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Τα ψηφιακά πώς θα την προστατεύσουν. Ιδιαίτερα στις επιγραμμικές πωλήσει που μπορεί να έχουμε πλαστά προϊόντα ή κατώτερης ποιότητας. Στην πράξη, στην ενιαία αγορά αυτοί οι κανόνες πώς διέπουν τα προϊόντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι του παραδοσιακού. Ευχαριστώ κύριος ε, Μπομπάχ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Μπρετό. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είπατε πόσο σημαντικά είναι τα ψηφιακά και τα δεδομένα στις κοινωνίες μας. Άρα αυτό συνδέεται με την τεχνολογία ε, και την αυτονομία τους της τεχνολογίας και των υποδομών για να έχουμε την κυριαρχία μας στα δεδομένα, άρα την κυριαρχία μας σκέτο και να μην ε, ε, υποκύπτουμε σε εξωτερικούς εκβιασμούς ή απόπειρε αποσταθεροποίηση. Σήμερα δεν είμαστε σε θέση να έχουμε αυτή την αυτονομία. Τα υποβρύχια, ας πούμε, καλώδια από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τα όσα αποκάλυψε το 2013 ο κύριος Σνόντεν, ε, εκεί σε αυτά τα ε, καλώδια γίνεται κατασκοπία βιομηχανική και, και ηλεκτρονική. Τι, έχετε μια, καμιά στρατηγική γι' αυτό για να μην επαναληφθεί. Επίσης για τις στρατηγικές μας εταιρείες ε, Alcatel Submarine Network ή Nokia πώς θα προστατευτούν από τα αρπακτικά από κάποιες ε, εξωτερικές εταιρείες. Επίσης θα ανοίξετε στην Ευρώπη data center όχι στη Silicon Valley, εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλέγκο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε ότι έχουμε τώρα μια νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό και διαπιστώσαμε ότι για το πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης ε, διαπιστώνουμε μειώσεις και περικοπές. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα ψηφιακή εποχή. Χωρίς ε, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους δεν μπορούμε να σταθούμε ανταγωνιστικά απέναντι στους κολοσσούς ε, αυτούς της ψηφιακές εταιρείες. Ε, η Ευρώπη έχει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στη ρομποτική επίσης. Σας ερωτώ λοιπόν, από τη μια έχουμε λιγότερη χρηματοδότηση και από την άλλη προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη ε, της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Με ευθύνη, με ευφύεια, αλλά και τεχνολογική αριστεία. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Τούν. Thank you. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τελειώνει αυτή η συνεδρίαση και επ' ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι η εμπειρία σας, η γνώση σας και το πάθος σας για την ενιαία αγορά είναι πραγματικά για μας πολύτιμα. Και αυτή η Λευκή Πίπλος για την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει επίσης ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ ε, καλά τα επόμενα χρόνια. Αλλά, αλλά στην ανακοίνωση για τη διαμόρφωση ε, του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, για μένα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που λείπει και αναφέρομαι στο γεωγραφικό αποκλεισμό, geo-blocking. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, είναι απρόθυμη να καταθέσει πρόταση για να αναθεωρηθεί αυτός ο κανονισμός, γιατί αν ισχύει αυτό είμαι βαθύτατα απογοητευμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Έχει πει μέχρι τις 31 Μαρτίου για αυτό το θέμα. Ο υφιστάμενος κανονισμός, θα γνωρίζετε σίγουρα, δεν βοηθάει τους καταναλωτές ε, να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Γι' αυτό θέλω να εξασφαλίσω ότι έχετε την πρόθεση να αλλάξετε την κατάσταση αυτή και μάλιστα επιγόντως. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι η δική μας πολιτική ομάδα παραδοσιακά επιθυμεί μια εσωτερική αγορά χωρίς ε, εσωτερικά σύνορα και μεγαλύτερη διάνοιξη της αγοράς προς τα έξω, εξαγωγική αγορά. Ε, ε, η στρατηγική για τα δεδομένα λέει ότι περισσότερα δεδομένα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κυκλοφορούν. Δεν φοβάστε διεθνείς αντιδράσεις Πώς θα βρείτε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανοιχτή και την κλειστή ε, κυκλοφορία και ροή δεδομένων ε, Ευρώπης Αμερικής. Ευχαριστώ. Έχετε πέντε λεπτά κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε και για τα καταληκτικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ. Για όλα, για όλα πέντε λεπτά. Ε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που είναι σε συζήτηση, οπότε θα πρέπει να ξαναέρθω να σας δω όλους μαζί έναν έναν για να μπορέσουμε να τα πούμε καλύτερα. Μην φοβάστε. Θα τα ξαναπούμε, μια που είναι τόσο ευχάριστο. Και απόψε είπαμε στο που καταλήγουν οι προσπαθίες μας. Είπαμε για τη Γενική Διεύθυνση Connect. Είναι πρώτο πρώτο το θέμα της χρηματοδότησης, το μήνυμα ελήφθη και προσέχουμε τη σχετική αλυσίδα αξίας. Κρυπτολογία και κβαντική τεχνολογία. Προσπαθούμε λοιπόν σιγά σιγά να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τώρα για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, το θέμα ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Όχι, δεν το ξεχάσαμε. Είναι προτεραιότητά μου. Και θα κάνουμε αυτό για το οποίο δεσμευθήκαμε. Και θα τα ξαναπούμε, αλλά δεν έχω αλλάξει γραμμή πλεύσης τώρα. Ένα θεματάκι που θέλω να σας πω για τις εφαρμογές ψηλού κινδύνου γίνανε οι προτάσεις αλλά και πρέπει να γίνονται οι διαβουλεύσεις και μεταξύ μας να καταλήξουμε ποιες είναι οι, μεν και ποιες οι δε εφαρμογές του υψηλού ρίσκου ή όχι. Είπαμε για τα παιχνίδια, για τα παιδιά, ναι, είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να υπάρχει η νομοθεσία για ευθύνη και ασφάλεια. Επίσης, μιλήσατε για αυτονομία στρατηγική για τα δίκτυα. Μα σε κάθε επιχείρηση. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και δεκαετία ήμουνα στις λεπικοινωνίες και είχαμε σχετικές δυσκολίες. Εγώ θεώρησα ότι ήταν στρατηγικό και εκτιμένο για την Ευρώπη η πολιτική για το προσωπικό. Και έχουμε σήμερα ένα ολόκληρο στόλο, ο πιο αποδοτικός. Είναι θέμα κυριαρχίας της ε, Ευρώπης. Οπότε σας είπα ότι αυτό ξέρω. Οπότε έτσι γίνεται με αυτά τα βιομηχανικά δεδομένα όσον αφορά την ε, αποθήκευσή τους, την επεξεργασία τους αυτά θα καταφέρουμε τη στρατηγική μας. Βεβαίως και θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του ΠΟΕ. Έχουμε τους εταίρους μας, αλλά έχουμε και τους κανόνες μας που θα πρέπει ξεκάθαρα να τους εφαρμόζουμε. Να ισχύουν για όλους και όσον αφορά τις ισχύωσες συμφωνίες χωρίς προστατευτισμό. Γιατί υπάρχουν Ε, όπως είπατε για το 5G κύριε Μπελαμή έχετε δίκιο υπάρχουν κάποια κριτήρια για το αν κάποιος πάροχος είναι υψηλού κινδύνου ή όχι και αν χρήζει όχι προστασίας και αν το λέει ο νόμος αυτός αποκλείεται άλλα στην επικοινωνία, άλλα στην βιομηχανία για τις εφαρμογές Άρα, θα πρέπει για τον ανταγωνισμό να εφαρμόζονται οι κανόνες. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη την εξέλιξη του τοπίου. Την εξέλιξη στα ψηφιακά. Αυτά που είπαμε σήμερα. Πάρα πολλά είπατε, πολύ για τις ΜΜΕ. Τα εξηγήσαμε. Ναι, όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση. και επομένως έτσι θα πρέπει να γίνει η διακυβέρνηση να καταπολεμηθούν όντως τα προϊόντα της παραποίησης ό,τι προϊόν είναι παράνομο τέλος πάντων οπότε αυτό θα το αναλάβουμε με την εκτονιστέρων νομοθεσία είναι στο χαρτοφυλάκιό μου και αυτή την αρμοδιότητα θα την αξιοποιήσω αυτά κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε ως απαντήσεις και ως συμπεράσματα. Μπουσόι. σας ευχαριστούμε πολύ εμείς. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Σήμερα μας παρουσιάσατε τις ε, προτεραιότητες σας και για αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα όσον αφορά τα ψηφιακά. Είναι βασικό αυτό για την Ευρώπη, για την βιομηχανία και έτσι θα πρέπει να προβλέψουμε και νομοθετικά, ούτω ώστε όλοι μαζί, κρατημέλη, επιτροπή και εμείς, να βοηθήσουμε για, για ανταγωνιστικότητα και άρα περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα βήματα για αυτή την ψηφιακή, την αλλαγή αυτήν, γιατί μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες ευκαιρίες και όσο γίνεται λιγότερους κινδύνους. Ευχαριστώ.